Right. Πάμε, ας ξεκινήσουμε το, το απόγευμά μας, όπως είπα το πρωί. Περιμέναμε και πήραμε και μια επιστολή από την Κορεπέρ, συμφωνώντας για τη συμφωνία για το ΣΕΠ. Και τώρα πρέπει να περάσουμε και στην επίσημη διαδικασία διαβούλευσης. Εν πάση περιπτώσει έχουμε το, την επιστολή αυτή και βάσει του άρθρου 70 παράγραφος 3 θα πρέπει να το να ζητήσω αν έχετε αντιρρήσεις προτού ε, παραπέμψουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, συγχαίρω την κυρία Σάια, την εισηγήτρια, ξέρω δεν μπορούσε να είναι παρούσα, αλλά έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς αυτό το θέμα Θέλω να την ευχαριστήσω. Δεν ήταν πάντα εύκολο να βρούμε κάποιον για να προεδρεύσει στον τριγωνικό διάλογο. Εγώ χρειάστηκε να την αντικαταστήσω κάποιες στιγμές. Εν πάση περιπτώσει τα κατάφερα μετά από πολλές από αυτές τις συνεδριάσεις που προείδρευσε. Νομίζω ότι καταφέραμε να συμπληρώσουμε αυτή τη διαδικασία υπό πολωνική προεδρία. Εξακολουθούμε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε βέβαια την κρίση του ευρώ και όπως σας είπα σήμερα το πρωί αυτό καταδεικνύει ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν με μεγάλη ευσυνειδησία να εργάζονται για να βελτιώσουν την εσωτερική αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με το ευρώ στον πυρήνα αυτών των υπηρεσιών. Είναι σημαντικό το θέμα λοιπόν της εμπιστοσύνης στο ευρώ και πιστεύω ότι όλα αυτά θα είναι πολύ θετικά για τους ε, επιχειρηματίες και τους καταναλωτές. Ζωάν Πολ, θες να πεις κάτι? Όχι? Μα πρέπει να ξεκινήσουμε με σένα. Δεν έχω καμία αντίρρηση, λέει ο Ζωάν Ευχαριστούμε. Είναι από τα πρώτα θέματα που μας απασχόλησαν μαζί τους δυο μας την τελευταία θητεία και πολύ χαίρομαι που όλα έχουν φτάσει πια στην εκπλήρωσή τους, στην κατάληξη της διαδικασίας. Πάμε στο σημείο 10 λοιπόν και την έκθεση ε, την ετήσια έκθεση μεγέθυνσης 2012 και τώρα ο Ζωάν Πολ είναι πράγματι ο εισηγητής για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προηγουμένως, σας υπενθυμίζω ότι ήμουνα σε μια στρογγυλή τράπεζα το μεσημέρι στην οποία συμμετέσχα και μου δώσανε ένα μήνυμα λέγοντας ότι η δημοκρατία επιβάλλεται, δεν είναι κάτι το οποίο το ζητάει κανείς. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για την έκθεση, για την ετήσια έκθεση μεγέθησης μου λέτε ότι αυτό είναι κάπως παράξενο, γιατί αυτό είναι μια συνηθισμένη άσκηση στην οποία υποβάλλεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φέτος είναι μια ευκαιρία για μας <clears throat> να καταδείξουμε τη θέληση του Κοινοβουλίου να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στον δημοκρατικό έλεγχο για τις οικονομικές πτυχές της ολοκλήρωσης στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν είχε την καλοσύνη να μας δώσει την έκθεσή της νωρίτερα από ότι προβλεπόταν. Έχουμε ήδη εργαστεί με όλους τους σκιώδεις εισηγητές γιατί εγώ κατέθεσα την έκθεσή μου στις 16 του μηνός και συζητάμε για πρώτη, συζητήσαμε για πρώτη φορά τις 19 του μηνός. Για την ουσία λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω μακρά σχόλια, βρίσκεται στο σχέδιο έκθεση το οποίο εγώ κατέθεσα, το σχέδιο έκθεση, το οποίο θα τροποποιηθεί βέβαια από τη στιγμή που η ΜΕΝ και η ΔΕ θα έχουν διατυπώσει τις τροπολογίες και τις προτάσεις τους. Επί της ουσίας του θέματος, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει η Κομισιόν είναι αρκετά λογικό και μπορούμε πολύ εύκολα να το αποδεχτούμε. Μια άλλη πτυχή όμως θέλω να θίξω, για την οποία συζητήσαμε και με τους χειώδεις ότι θα πρέπει να βρούμε πώς αυτή η έκθεση του Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης μπορεί να εγγραφεί σε αυτή τη νέα δομή που προκύπτει από την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στην Επιτροπή Απασχόλησης υπάρχει μια διαδικασία σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές, βάσει της οποίας διαδικασίας η Κομισιόν, η Επιτροπή μας μάλλον και η Πρόεδρός μας επέτυχε να επιτύχουμε ένα σχήμα ιονής συναπόφασης. Βέβαια, η κατάσταση αυτή δεν είναι ακριβώς η ίδια για το τρέχον θέμα, γιατί για τις κατευθυντήριες γραμμές απασχόληση υπάρχει μια σαφή συμφωνία, ενώ για την ανάπτυξη είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι θα βρούμε το δρόμο μας περπατώντας και κινούμενοι. Ελπίζω κατά τη διάρκεια αυτή τη συζήτηση θα έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου κατά τρόπο ώστε να είναι πιο συνεκτική και η δράση μα μαζί με τα αιτήματα που έχουμε διατυπώσει, τα θεμητά μα αιτήματα σε σχέση με την ύπαρξη και τη λήψη υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου για θέματα τα οποία είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα πια και τα οποία απαιτούν δημοκρατικό έλεγχο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να προωθήσουμε αυτή την κατάσταση. Είναι γεγονό ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια εξέταση αυτού του φακέλου σαν να επρόκειτο πλήρω για διαδικασία συναπόφαση. Αυτό θα ήταν υπερβολικό από τη δική μου πλευρά, πολύ βεβαιασμένο και θα μα ε, παρουσίαζε σαν να τα είχαμε παίξει. Όπω λένε οι νέοι, ότι είχαμε ξεφύγει από τα όρια και αυτό δεν θα οδηγούσε σε τίποτα, θα ήταν χαμένο κόπος. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα άλλο τρόπο, αλλά αυτό αξίζει να το συζητήσουμε προηγουμένω, να βρούμε ένα άλλο τρόπο, ενδεχομένω να τολμήσουμε, και το λέω σαφώ να τολμήσουμε να υποβάλουμε σαφείς προτάσει, οι οποίε θα είναι ισοδύναμε με τροπολογίε <clears throat> στο τέλο τη έκθεση αυτή, η οποία μπορεί να παρουσιαστεί ω ένα σύνολο προτάσεων από τη μεριά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις οποίες το Κοινοβούλιο θα ήθελε να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της εκπόνησης των προοπτικών για την ανάπτυξη. Αυτή είναι λοιπόν η μέθοδος που σας προτείνω. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τους σκιώδεις εισηγητές. Έχουμε και μία ε, συνεδρία εργασία για τα θέματα αυτά. Πιστεύω όμως ότι το ύφο της σημερινής συνεδρίασης, της σημερινής συζήτησης μάλλον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο επωφελώς για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να εκφράσουμε τη θέση και τη θέληση του Κοινοβουλίου και να εξασφαλίσουμε στο μέλλον μια πιο άμεση συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου, Κομισιών και Κοινοβουλίου, η οποία θα μπορούσε να πλησιάσει την συναπόφαση και να πάρει αυτή τη μορφή μετά από κάποια μεταγενέστερη μεταρρύθμιση των συνδικών. Το Κοινοβούλιο λένε πολλοί ότι δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει με τέτοιο ε, προορατικό τρόπο στα θέματα αυτά. Εγώ νομίζω όμως ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο, να έχει μια ταχεία αντίδραση στα θέματα αυτά. Είδαμε σε σημαντικά θέματα πολύ πριν από τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν όλα βέβαια την ίδια πολιτική παράταξη. Ανήκουν στην ίδια παράταξη, το Κοινοβούλιο είχε καταφέρει να έχει επιτύχει μια συμφωνία. Δεν είναι θέμα λοιπόν ταχεία αντίδραση, είναι θέμα σωστή εργασία, σωστή οργάνωση των εργασιών μα και από τη στιγμή που μπορούμε να σεβαστούμε τα χρονοδιαγράμματα, μπορούμε να οργανωθούμε και να εργαστούμε με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τηρήσουμε τις προθεσμίες και αυτή τη φορά η ημερομηνία που κατέθεσε το σχέδιό της η Κομισιόν μας δίνει ένα χρονικό διάστημα επαρκές αν εργαστούμε με μεγάλη ταχύτητα ε, εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε να προωθήσουμε τα πράγματα δεν μιλάω για τον εαυτό μιλάω για όλους μας αν το Κοινοβούλιο λοιπόν θέλει να εξασφαλίσει ότι θα έχει τις εξουσίες που είναι η βάση του δημοκρατικού ελέγχου, θα πρέπει να είναι σε θέση να πράξει τα απαραίτητα και για να αντιδράσει ταχαίως και επίσης να μπορέσει να διεκδικήσει και να κατακτήσει τις εξουσίες του. Σας ευχαριστώ. Ε, thank you. Σας ευχαριστούμε, Περβάνς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για αυτή την πολύ καλή βάση για τις συζητήσεις μας. Είναι η δεύτερη φορά που πρέπει να αποφανθούμε για την ετήσια έκθεση ανάπτυξη. Είναι η δεύτερη φορά που μα υποβάλλει αυτό το έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε ακόμα στη φάση τη ε, προετοιμασία. Τέλο πάντων, ευχαριστούμε που τέλου αποδέχεστε την ιδέα ότι το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει καθήκοντα συναπόφαση. Είναι όμως και η πρώτη φορά που παρεμβαίνουμε για την ετήσια αυτή έκθεση ανάπτυξης, όπου εκ νέου βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν ότι το φύλλο πορεία του για τι οικονομικέ πολιτικέ ω κείμενο δεν έχει υπάρξει αντικείμενο καμιά συζήτηση. Σε κανένα κοινοβούλιο, σε κανένα μέρο του κόσμου. Και αυτό ονομάζεται σύμφωνο Europlus. Αν δείτε το σχέδιο συνθήκης που προσωρινά αποφασίσαμε να το αποκαλούμε συμφωνία η μία, είναι σύμφωνο Europlus και αναφέρεται αυτό τουλάχιστον τρεις φορές. Ε, είναι μια συμφωνία διακυβερνητική, αλλά δεν έχει συζητηθεί σε κανένα κοινοβούλιο, δεν έχει περάσει από καμία διαβούλευση, καμία κύρωση κοινοβουλευτική. Αυτό λοιπόν που επανεισάγουμε είναι μια διαδικασία όπου τα κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν. Βέβαια, Εμείς ε, θα υψώσουμε τη φωνή μας για να πούμε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη στρατηγική, την εξέταση της στρατηγικής ανάπτυξης, κάτι που επιλέξαμε να ονομάζουμε αιτήσιου προσανατολισμού ανάπτυξη. Όμω εντωμεταξύ αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων προχωρούν στην εξέταση ενό κειμένου όπου ουσιαστικά μα τριμώξανε για να συμμετάσχουμε στην όλη διαδικασία. Και αυτό το σύμφωνο ονομάζεται γύρω πλάσιο τους διαπραγματευτές. Θα τους συναντήσουμε στο τέλος ε, της μενής μέρας και θα πρέπει να δούμε στην όλη συζήτηση αν το σύμφωνο αυτό μπορεί να ονομάζεται, μάλλον αυτή η συμφωνία μπορεί να ονομάζεται σύμφωνο Europlash. Δεν ξέρω κατά πόσον το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να συμμερίζεται αυτέ τι απόψει. Σα θυμίζω ότι όταν ήρθε ένα εκπρόσωπο τη Πολωνική Προεδρία ε, σε μια από τι ιστορικέ συνόδου που οργάνωσαν, όταν το ρωτήσαμε για το θέμα αυτό, μα είπε ότι ξεκάθαρα για εκείνον η ετήσια εξέταση ανάπτυξη πριν να καλύπτει και το σύμφωνο Europlus. Αυτό το λέω για το γενικότερο ε, τοπίο εντό το οποίο κινούμαστε. Τώρα, ε, η στατικική του εισηγητή ήταν να ετοιμάσει ένα σύντομο κείμενο με κάποια σοβαρά πολιτικά μηνύματα. Σας ευχαριστώ που έτσι εξετάσατε το θέμα. Αλλά καλά θα ήταν να υπάρχει και ένα παράρτημα όπου να λέμε συγκεκριμένα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τι θα σήμαινε να διορθωθεί το κείμενο ετήσιας έκθεσης για την ανάπτυξη. Τώρα προς το ίδιο το πολιτικό μήνυμα που θέλουμε να αποσταλεί μίλησα για τις αναφορές στο σύμφωνο Europlus. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Όταν εγκριθεί το κείμενο αυτό, η στιγμή θα είναι κέρια. Θα εκτελήσονται παράλληλα διαπραγματεύσεις για το υποσυζήτηση κείμενο ως προς τις προτεραιότητες που προτείνονται. Στο κείμενο δίνεται έμφαση προφανώς στο θέμα της διαχείρισης των κρατικών χρεών. Προφανώς σε σχέση με τι προτεραιότητε όπως τις ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι το ζήτημα της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε σαν αποτέλεσμα των υπόλοιπων συνιστοσών της στρατηγικής. Αλλά αυτό δεν είναι επικριτικό σχόλιο προς τον εισηγητή, αλλά από την δημοσιονομική από την αρχή μάλλον που καθορίζεται τη δημοσιονομική πειθαρχία χωρίς να πρικοδοτηθεί με τα μέσα που επιτρέπουν την πειθαρχία αυτή και τα μέσα που επιτρέπουν την ανάπτυξη επίσης. Χαίρομαι πάντω ιδιαίτερω για τις προτάσεις του εισηγητή. Ιδίω εκεί που αναφέρεται στην ανάγκη επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευση τη έρευνα της καινοτομία των υποδομών και τη ενέργεια, Νομίζω ότι ο άξονας αυτό είναι πρωταρχική σημασία. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια συμβαστική λύση πολύ ισχυρή. Θα πρέπει να είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηνύματα που θα περάσουν από την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Στην παράγραφο 9 για το θέμα της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της κατάστασης των τραπεζικών κεφαλαίων εδώ θα πρέπει να το δούμε και με τον κύριο Κάρας βεβαίως ποιο μήνυμα ακριβώ θέλουμε να αποστείλουμε αλλά Υπάρχει η χρονιά κίνηση το 2012 που είναι πολύ σημαντική διότι οι τράπεζες προσπαθούν να προλάβουν την παρέμβαση που επίκειται, αλλά υπάρχει και η αξιολόγηση των κρατικών ε, χρεών εν Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι μήνυμα θα περάσει με αυτό το σημείο. Στο 10, η περίφημη μνήμα στι διευθυντικέ μεταρρυθμίσει. Δεν έχω καμία αντίρρηση να μιλήσουμε για όποια διαφορετική μεταρρύθμιση θέλετε. Όμω, καλό είναι πρώτα να ορίσουμε τι εννοούμε με το διαφορετική μεταρρύθμιση. Διότι διαφορετική μεταρρύθμιση που απλώ οδηγεί σε την αριθμική προσαρμογή των μισθών ή σε μείωση των συντάξεων, αυτό δεν μου φαίνεται ότι είναι ένα σημείο στο οποίο μπορούμε όλοι να αποσπάσουμε συνένεση και μάλιστα με τρόπο εύκολο. Η αναφορά αυτή γίνεται και στην ενδέκατη παράγραφο. Εκεί η διατύπωση κάπως με δυσκολεύει. Τέλο πάντων, δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλώς να ευχαριστήσω ξανά τον εισηγητή για την προθυμία του, τη συνεργασία του και για το χρονοδιάγραμμα και για την προσέγγιση του στις διαπραγματευτικές μεθόδους που ακολουθεί ως προς το Συμβούλιο. Το οποίο, όπως είπα, δεν είναι ξεκάθαρο. Είμαστε σε μια φάση που αυτό το σημείο θα τραβήξει όλη την προσοχή. Θα βρεθεί στην καρδιά των διαπραγματεύσεων. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχει νόημα όλη αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει να συνδυάσουμε δύο διαφορετικά είδη εργαλείων. Θα πρέπει να τα διαρθρώσουμε. Τα δύο αυτά εργαλεία, πρέπει να τα θυμίσω, είναι από τη μια η στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, που δεν πρέπει να παραμείνει καινογράμμα, αλλά θα πρέπει να μεταφραστεί σε υλική πραγματικότητα, ιδίω τη στιγμή που θα καθορίσουμε τι δημοσιονομικέ στρατηγικέ των κρατών μελών από τη μία, και από την άλλη το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Και αυτό με τη σειρά του θα πρέπει να μεταφραστεί σε προγράμματα σταθερότητα και σύγκληση των κρατών μελών. Προτού καλυφθεί στις ειδικέ αναχώρα τάσεις. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε, Σιλβί. Ευχαριστώ, Σάρον. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Πραγματικά βρισκόμαστε στα πλαίσια μιας διαδικασίας εξελισσόμενης. Το ΣΥΚΣΠΑΚ, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, τώρα συνεχίζουμε με τη συνθήκη. Είναι πάντοτε λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς μπορεί να απονομονώσει χρονικά αυτά τις ε, αλληλένδετες φάσεις της ίδιας διαδικασίας. Με την ε, Περβάνη θα συμφωνήσω στο εξής ότι υπάρχει κατάφορη έλλειψη δημοκρατικής εξέτασης του συμφώνου Europlus. Ε, υπάρχει, εδώ έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με πολιτικές δηλώσεις, αλλά ήδη αναφέρονται και γίνονται υπενιγμοί για την νομοθεσία. Συνθήκη αναφέρθηκε, θα βρεθεί στην κορυφή της νομοθεσίας, ακόμη και αν είναι διεθνής αυτή η συνθήκη, και αυτό με ενοχλεί βαθύτατα. Διότι βρίσκω ότι εδώ υπάρχει οπισθοδρόμηση. Ακόμη, εάν σκεφτούμε τι διαδικασία ακολουθήθηκε για τη στρατηγική του 2020. Και η στρατηγική αυτή δεν αναφέρεται καν στι πρόσφατε δηλώσει. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει κάποια διαφορά, κάποια κόποση, διότι φαίνεται ότι με την επιδίωξη του τέλειου τελικά πετάμε μαζί αυτό που ήδη είχε επιτευχθεί ως αποτέλεσμα. Εδώ τώρα θα πρέπει να θέσουμε σωστά τι προτεραιότητέ μα. Ε, λέμε στο κείμενο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει προτεραιότητε, τι οποίε εγώ δεν έχω να τι αμφισβητήσω, δεν έχω κάτι εναντίον του. Όμω, όταν μιλάμε για τη στρατηγική του 2020, δεν τι ξαναβρίσκουμε. Επίση, θα συμφωνήσω με το Ζαν Πολ ότι πρέπει εδώ να υπάρξει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια, λεπτομερή ανάλυση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι εδώ σαφώς χρειάζεται συμβολή και του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν περισσότερο να σκεφτούμε τον κίνδυνο επικάλυψη των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, να παραμεριστούν οι σημαντικέ συζητήσει κοινωνικού περιεχομένου για τη φορολογία εκτό του θεσμικού πλαισίου και κυρίως να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το κείμενο αυτό σε λογικές διαστάσεις. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την περσινή έκθεση έχει αλλάξει κάπως την, το πνεύμα υπό το οποίο προσεγγίζει το θέμα αυτό, αλλά αυτή είναι οι βάση της συζήτησης, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περαιτέρω. Ο Φιλίπ, σε ευχαριστώ Sharon. Ευχαριστώ, Ζαν Πολ, και καλημέρα. Πρέπει να αναφερθώ στον Κριστιαν σε σένα. Ωραία, στον Ζαν Πολ μιλάω τώρα. Για την έκθεση αυτή, καταρχήν σε σχέση με τη δομή της. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο έκανε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. Νομίζω ότι αυτά που είπε η Σιλβή είναι ουσιαστικά και η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θεώρησε ότι υπάρχουν τρία-τέσσερα σημεία στα οποία μπορεί να τροποποιηθεί η ετήσια έκθεση ανάπτυξης. Είναι πολύ καλά διαφρομένη λοιπόν η γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε και εμείς μια τέτοια δομή για να είναι σαφές και το μήνυμα το οποίο θα δώσουμε στο Λομπέλι. Αυτό το πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι μπορεί να έχει περισσότερες αποχρώσεις αυτή η διατύπωση τώρα, αλλά έχει λιγότερη συνακτικότητα. Υπάρχουν πολλοί στην Κομισιόν που του ενδιαφέρει η αναδιανομή, η αντιμετώπιση της ένδυας. Αυτό είναι θετικό από την άλλη μεριά. Παραμένει το μήνυμα της μονομανίας με την ε, λιτότητα στον προϋπολογισμό και τις περικοπές και δεν βλέπουμε σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να είναι σημαντό με μια πολιτική αναδιανομή. Αυτό είναι το πρώτο σημείο για το οποίο θα πρέπει εμεί να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ισορροπία. Και εδώ συμφωνώ με τη Σιλβή σε σχέση με τη στρατηγική Ευρωπαϊκή 2020. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση στα πλαίσια του SIXPAC των έξι νομοθετημάτων με στόχο να γίνει πιο δεσμευτικό το σύνολο των στόχων της στρατηγικής 2020 και εδώ πάλι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δούμε την αναγκαιότητα της στρατηγικής αυτής. Αν είναι έτσι λοιπόν, θα πρέπει η Κομισιόν και στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης προόδου σαφές <clears throat> ότι δεν πρέπει να υπάρχει μονάχα σαν πρώτη, σαν δεύτερη, σαν τρίτη σύσταση λιτότητα και ίσως κάποια υποσημείωση που να λέει ναι υπάρχει και κάτι που λέγεται στόχος της Ευρώπης 2020. Αλλά αντίθετα θα υπάρχει μια μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη λιτότητα του προπολογισμού και με μια όθηση προς τις επενδύσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δώσουμε λοιπόν στις συστάσεις μας. Για τα εγκάσια θέματα και πάλι, για μένα παραμένει το θέμα των μακροοικονομικών ανισομεριών που πρέπει να αναφερθούν και των αποτελεσμάτων των λεγόμενων spillover effects, δηλαδή των παραπλεύρων αποτελεσμάτων μπορεί να προκύψουν. Μια χώρα δηλαδή, που έχει προβλήματα μπορεί να προκαλέσει τέτοια αποτελέσματα και στις γειτονικές χώρες. Εδώ θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο εκπεφρασμένοι από ό,τι λέει το κείμενο προς το παρόν. Εμένα μου φαίνεται ότι κάπου η λεγόμενη Ordnungspolitik, η πολιτική του να βάζουμε τα πράγματα σε κουτάκια, κάπου το έχει σφραγίσει ιδιαίτερα το κείμενο αυτό. Στην παράγραφο 6 λέμε η έξοδος από την κρίση για τα κράτη-μέλη εξαρτάται από την ικανότητά τους να ανταποκριθούν με αποφασιστικό τρόπο στην κρίση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν οι μακροοικονομικές ανισομέρειες που ανέφερα προηγουμένως, στο να μπορέσουμε να ελέγξουμε και πάλι τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Και πάλι δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι το σύνολο θέμα τη λιτότητα του προπολογισμού είναι δευτερεύον, αλλά ούτε είναι και πανάκια. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν και πολλά άλλα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό είναι ένα γεγονό. Δεν είναι απλώ μια σχετικοποίηση. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του προπολογισμού χωρί να λύσουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να υπενθυμίσω και στο ΣΥΚΣΠΑΚ το είχαμε πει προηγουμένω ότι οι δημόσιε δαπάνε δεν μπορούν να αυξάνονται ταχύτερα από τον προσδοκόμενο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ εκτός εάν υπάρχει κάποια μορφή αντιστάθμισης η οποία είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Ούτε αυτό πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Αν πούμε απλώς ότι οι, οι δεν προχωρούν πιο γρήγορα από την αύξηση του ΑΕΠ, αυτό το παρασιωπούμε. Παράγραφος 10. Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει τόνωση της ε, εσωτερικής ζήτησης και πάλι πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τα ελλείμματα αλλά και τα υπερβολικά πλεονάσματα. Και αυτό είναι αυτό το οποίο θέλω να τονίσω. Η Περβάνς γνωρίζει ότι το θέμα των διαφθορτικών αλλαγών είναι κάτι το οποίο έχει δηλητηριαστεί αυτή η έννοια. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για την ε, εργασία μονάχα σαν να είναι θέμα κατανομής εργασιών θα πρέπει η Κομισιόν να κάνει το δικό τη καθήκον και εμεί το δικό μα καθήκον και εγώ έχω κάποιε τροπολογίε οι οποίε είναι επικοδομητικέ ελπίζω. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Χουντή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα μας έδωσε μια βάση για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Να μου επιτρέψετε να πω όμως ότι το πρόβλημα για μας δεν είναι θέμα χρόνου ή πιο έγκαιρης κατάθεσης από την πλευρά της Επιτροπής της Ετήσιας Επισκόπησης, που είναι κάτι θετικό, εν πάση περιπτώσει, ούτε όμως είναι πρόβλημα απλά δημοκρατικής νομιμοποίησης. Σύμφωνοι, να διεκδικήσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην περίπτωση που υπάρχουν και αναθεώρηση των συνθήκων αυτό να είναι και θεσμικά κατοχυρωμένο. Λέω, it's a noise. Ε, Είπα ότι το κύριο πρόβλημα δεν είναι το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης και σωστά να διεκδικήσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως εισηγείται η έκθεση σε περίπτωση αλλαγής συνθήκων να έχουμε πιο ουσιαστικό ρόλο σύμφωνοι σε αυτό. Όμως το θέμα είναι κατεξοχήν πολιτικό και με αυτή την έννοια διαβάζοντας και το κείμενο της ετήσιας επισκόπησης της Κομισιόν διακρίνω ότι ο εισηγητής ταυτίζεται σχεδόν με το πνεύμα και τις κατευθύνσεις της ετήσιας επισκόπησης. Και τώρα τι έχουμε, μια ετήσια επισκόπηση για το 2012 που είναι στην ίδια κατεύθυνση που ήταν και η ετήσια επισκόπηση του 2011 και αναφέρομαι στο κείμενο της Κομισιόν αλλά που προθεί ή θέλει να προωθήσει τις ίδιες πολιτικές με πιο βίαιο κατά την άποψή μας και πιο εσπευμένο τρόπο την ίδια ώρα που ακούμε για νέα συνθήκη και ούτω καθεξής, αυτή το κείμενο της Κομισιόν ουσιαστικά πάει προς την ίδια κατεύθυνση. Βλέπει σαν του προβλήματος της κρίσης την ένταση των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων. Αυτό το μοντέλο έχει αποδειχτεί πια και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το παραδέχονται ότι οδηγεί στην ύφεση, οδηγεί σε μεγάλες κοινωνικές ανισότητες κατεδαφίζονται κοινωνικές κατακτήσεις, δεν έχει οικονομική αποτελεσματικότητα, δεν βγάζει κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, δεν φαίνεται να εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εφόσον λοιπόν αυτό το κείμενο της ετήσιας επισκόπησης αποτελέσει και θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση του δεύτερου ευρωπαϊκού εξαμήνου, για το οποίο κουβεντιάσαμε, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα για να αντιμετωπίσεις την κρίση με βάση τις ίδιες λογικές. Δεν θέλω να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά γιατί από τα όσα είπα πέρα από την προσπάθεια να διεκδικήσουμε έναν πιο ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συμφωνούμε με τις βασικές κατευθύνσεις που κινείται η έκθεση εφόσον και στο βαθμό εναρμονίζεται, σε όποιο βαθμό εναρμονίζεται με την ε, έκθεση που κατέθεσε η Κομισιόν για την ετήσια επισκόπηση. Επομένως διαφωνούμε με την ουσία του κειμένου, όχι στο συγκεκριμένο θέμα όσο αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια της προσπάθειάς μας με τροπολογίες θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, Νίκο. Αντυχεί πολύ, έχει αντίχηση εδώ πέρα και γίνεται φασαρία εύκολα. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να κάνουν περισσότερη ησυχία. Συγγνώμη, έβλεπα TV και ο Ντέρεκ θα μιλήσει τώρα, έτσι. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Γκοζές, για την έκθεσή του που είναι προσεκτικά συνταγμένη. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η μορφή του κειμένου μετά τις αλλαγές και τη διαδικασία τη συμβιβαστική, αλλά στην παρούσα μορφή μπορούμε να υποστηρίξουμε το πνεύμα και την διατύπωση. Η αυτή η επισκόπηση του 2012 ξεκινά το δεύτερο ευρωπαϊκό εξάμεινο της οικονομικής διακυβερνήσεως, καθορίζει τις προτεραιότητες για τη δράση και σε επίπεδο εθνικό και σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιε θα πρέπει να είναι οι βασικέ προτεραιότητε. Αν με ρωτάτε ποια βασική προτεραιότητα θα ήθελα, θα ήθελα να παραθέσω αυτό που είπαν ο Κέννεντι και ο Ρίγκα. Ε, ότι όταν ε, έχει ε, παλήρια και ανεβαίνει το νερό, σηκώνει και το πλοίο σου. Ε, αυτό θα ήταν κάτι υποφελέ, ε, ανάπτυξη ήταν υποφελή για την οικονομία. Θα έπρεπε να δούμε τι γίνεται από την πλευρά τη της παροχή. Να υπάρχει ευκολία να παρέχονται τα αγαθά και υπηρεσίε από τον κόσμο. Οπότε θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, λιγότερη ρύθμιση και να απελευθερωθούν οι αγορές. Μπορεί να ακούγεται παράλογο ε, για τον εισηγητή. Χρειαζόμαστε περισσότερα, περισσότερη οικονομία του Ρίγκαν για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση ε, στην Ευρωζώνη. Η έκθεση ως έχει τώρα, αν εξαρτιόταν από μένα, θα μπορούσε να ε, υιοθετηθεί και ως έχει, αλλά εντάξει θα προταθούν κάποιες αλλαγές. Η Ελίσσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επαναλάβω όσα ήδη υπόθηκαν, Απλώ οι βασικέ μου παρατηρήσει είναι οι εξή. Θεωρώ ότι η έκθεση έχει θετικές πτυχέ. και νομίζω ότι με τρόπο ενδιαφέροντα που βεβαίω μπορεί να βελτιωθεί περιττέρω, καλύπτει το ρόλο του Κοινοβουλίου και πώς μπορεί να ευλεχθεί το Κοινοβούλιο στην όλη διαδικασία ω προ το περιεχόμενο. Νομίζω όταν ε, μιλάμε για το Sixpack, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν είναι ότι δεν υπήρχε πρόγραμμα προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη, για την καινοτομία και τη σύγκληση. Έχουμε τώρα παρά την έλλειψη απόλυτης συνένεσης σε μία τέλο πάντων συμφωνία. Αλλά λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα πρόγραμμα προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη, ώστε να αντισταθμίσουμε αυτό που δεν καλύπτωταν από το six Το six επικεντρωνόταν υπερβολικά στην πειθαρχία, την, ε, τον έλεγχο, τις κυρώσεις. Δεν νομίζω ότι τώρα πρέπει να επαναλάβουμε τα ίδια όταν αναλύσουμε την ε, ετήσια μελέτη ανάπτυξης, δεν νομίζω ότι να επαναλάβουμε στοιχεία τα οποία ήδη τα έχουμε καλύψει στο Sixpack. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να θέσουμε μια ατζέντα για την ανάπτυξη και την ε, σύγκληση. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν έμφαση στα στοιχεία αυτά. κάτι που θα πρέπει να το δούμε και στο επίπεδο ορολογία, όπω στην παράγραφο 10. Λέγεται εκεί ότι υπάρχει ανησυχία γιατί πολλά κράτη-μέλη δεν αναπτύσσουν την παραγωγικότητά του. Μα αυτό είναι σχετικά περιθωριακό σε σχέση με τη συμφωνία επί τη αρχή για το ποιο θα είναι το κείμενο και η ουσία και θα πρέπει να είναι το κείμενο και η ουσία τη ετήσια έκθεση ανάπτυξη. Να δώσουμε λοιπόν μεγαλύτερη έμφαση στην ε, ανάπτυξη και την σύγκληση και όχι πάλι στην πειθαρχία. Επίσης, ελπίζω ο εισηγητής να με ακούει να ολοκληρώσει τη συζήτησή του. Συνάδελφοι, και πάλι, εάν μπορείτε να μην δυσκολεύετε τόσο τους ομιλητές, γιατί μετά θα έχουμε και τις ψηφοφορίες. Εάν μπορείτε λοιπόν τα πηγαδάκια Κύριε Γκοζές, να περιμένω ή να συνεχίσω. Καλώς. Θα ήθελα επίσης να βρίσκω, να έβρισκα στο κείμενο μια πιο συγκεκριμένη μνήμα για τη συνιστόσα των μακροοικονομικών ανισορροπιών από τα συστατικά του Δεν νομίζω ότι πρέπει τόση έμφαση να δοθεί στην διάσταση της πειθαρχία, αλλά ουσιώδες είναι να ενισχυθεί η συναστόσα των spillovers όπως λέγονται και του στοιχείου της σύγκλησης. Έπειτα, κατά τρίτο, νομίζω ότι στην 7η παράγραφο ήδη σχολιάστηκε από τον Φιλίπ η αναφορά στο συγκεκριμένο τεχνικό στοιχείο που θα πρέπει να υπάρχει για τον περιορισμό της αύξησης των δαπανών και το συσχετισμό με, το μεσοπρόθεσμο, με την αύξηση του μεσοπρόθεσμου ΑΕΠ, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ λεπτομερές στον σχεδιασμό και λείπει μια σειρά από αιτιολογήσεις εδώ. Θα μπορούσαν να προσθεθούν, να υπάρχουν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία. Τελευταία παρατήρηση στην ίδια κατεύθυνση, παράγραφος 11. Νομίζω ότι αναφορά στις μεταρρυθμίσεις της εργασιακής αγοράς. Για τους ίδιους λόγους και σε αυτό το πλαίσιο, με συγχωρείτε, υπάρχει κόσμος που μιλάει. Ο μόνος που θέλω να μιλάει εδώ και να ακούω τη φωνή του είναι η Ελίζα Φερέιρα και μετά η κυρία Χίμνερ. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω να διακόπτω και να ζητάω ησυχία. Θα καθυστερήσουν οι ψηφοφορίε. Μπορείτε λιγάκι να πειθαρχήσετε, εάν δεν θέλετε να καθυστερούμε. no Στην παράγραφο 11 έλεγα αντί να ζητάμε απλώς μεταρρυθμίσει στην εργασιακή αγορά και να μιλάμε για το επίπεδο της μισθοδοσίας, σημαντικό είναι εξίσου να αναφέρεται η ανάγκη να αυξήσουμε την επένδυση στην εκπαίδευση, τη στατηγική του 2020. Και έτσι να ενισχυθούν οι μισθοί. Ίσως έτσι να είναι δυνατόν να τους αυξήσουμε εφόσον θα μπορέσουμε να στηρίξουμε και την παραγωγικότητα, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού, πέραν των όσων έχουν υποθεί στα προηγούμενα κείμενα για τους μισθούς και την ε, ευελιξία που πρέπει να έχουν οι εργασιακές αγορές. Λοιπόν, ως προς το περιεχόμενο, η ετήσια έκθεση ανάπτυξης θα πρέπει να αντισταθμίσει την υπερβολικά περιοριστική ατζέντα που εγκρίναμε μέσω του Six Pack. Γι' αυτό άλλωστε ψήφισε αρνητικά και η ομάδα των σοσιαλιστών. Και επίσης θα πρέπει να προσθέσουμε κάποια στοιχεία από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, την ανάλυση των spillovers και ποιοι είναι οι όροι για την ε, ενίσχυση της ανάπτυξης. Τα τέταρτον, να ξαναδούμε στην 7η παράγραφο το θέμα του συσχετισμού μεταξύ των κρατικών δαπανών και την αύξηση του ΕΠ και τέλος, επαναλαμβάνω στην 11η παράγραφο, πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και όχι μόνο να επιμένουμε διαρκώς για την μείωση των μισθών. Το μήνυμα αυτό θα μπορούσε να περιέχεται να μην είναι τόσο ρητά διατυπωμένο. Ευχαριστώ, η Ευχαριστώ, Σάρων. Να σχολιάσω εν συντομία το σημείο 10 της εκθέσεως του Ζαν Πολ Γκοζές που αφορά σε θετικές αλλαγές. Πιστεύω ότι το εξάμεινο αυτό δεν αφορά μόνο τη δημοσιονομική πειθαρχία και τον πολιτικό συντονισμό, παρόλο που σημαντικά θέματα, αλλά είναι και σημαντικό μέσο που έχουμε στα χέρια μας να σπρώξουμε να γίνουν οι ε, διάφορες θετικές μεταρρυθμίσεις και θα ήταν χρήσιμο να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει κάποια επισκόπηση των διθωτικών ε, μεταρρυθμίσεων για να δούμε τι έχουν κάνει τα διάφορα κράτη-μέλη, τι κάνουν σε φασιστικές ε, αλλαγές και εκεί θα πρέπει τακτικά να παράγεται τέτοιο έγγραφο πιθανότατα ετήσια να γίνεται μια επισκόπηση του πώ προχωράνε στα διάφορα κράτη-μέλη ε, οι διαθωτικέ αλλαγέ. Ζαν Πολ, θε ξανά το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομο θα είμαι γιατί αλλιώ θα με πνίξουν αυτοί οι οποίοι αδειμονούν για την ψηφοφορία. Εγώ κατέγραψα όλα αυτά που είπαν και οι μεν και οι δε. Υπάρχουν δύο πτυχέ στο θέμα αυτό. Η πρώτη πτυχή είναι το θέμα του μηνύματος που θα πρέπει να δώσει το Κοινοβούλιο σε σχέση με την δική του αντίληψη για το πώς πρέπει να συμμετάσχει στη διαμόρφωση των μεγάλων κατευθυντηρίων γραμμών στα οικονομικά θέματα και από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα της ουσίας και εδώ κατέγραψε τις απόψεις των μεν και των δε. Προφανώς θα πρέπει να καταφύγουμε σε κάποιες συμβαστικές λύσεις γιατί σε πολλά θέματα αποκλίνουν σημαντικά οι θέσεις μας. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο είναι όμως να μπορέσει να βρει το ταχύτερο δυνατόν αυτές τις συμβαστικές λύσεις και να μπορέσει να συμπληρωθεί αυτή η κοινή έκθεση και να καταλήξει σε ένα σαφές μήνυμα για τα πιο ουσιώδη στοιχεία γιατί αυτό που χρειάζεται σήμερα δεν είναι να γράψουμε ένα, μια πραγματή πολυσέλιδη που θα μείνει στα ράφια αλλά να δώσουμε ένα σαφές και χμηρό μήνυμα το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί παρά τις διαφορές μας από όλο το Κοινοβούλιο και το οποίο θα καταδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε με ενεργό και δυναμικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Ευχαριστώ, πρόεδρος. <clears throat> Ευχαριστώ όλους. Ναι, πράγματι. Εδώ κρυώνω. Δεν ξέρω εσείς αν Η Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 12 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Αυτό είναι το μάξιμο που μπορούμε να πετύχουμε. 23 Ιανουαρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες, 24 θα ψηφίσουμε για να πάμε στην πρώτη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ λοιπόν. Και τώρα μπορούμε να πάμε στις ε, ψηφοφορίες. Και η πρώτη ψηφοφορία Μία δοκιμαστική ψηφοφορία πρώτα. Άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. Πατήστε το κουμπί που θέλετε. Δοκιμαστική ψηφοφορία είναι εξελίξη. Δοκιμαστική. 42 κάρτες, 43 κάρτες, 42, 41, κάποιος δεν ψήφισε, εσύ φταίς. Κάποιος δεν ε, πάτησε το κουμπί ακόμα. Δύο δεν πάτησαν το κουμπί. Τρεις δεν πάτησαν το κουμπί. Λέει πρώτος. Και τώρα έχουμε μία παραπάνω ψήφο από το ΕΛΚ. Ένας από το ΕΛΚ περισσεύει. Εντάξει. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. 36 ικανοποιημένοι βουλευτές. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία λίγη σιωπή. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Θέλετε το λόγο. Όλε, όλε. Αν ξεκινήσουμε, ήθελα να ρωτήσω αν ξεκινάμε την έκθεση για, το, για τα φορολογικά. Στη συνάντηση των συντονιστών αποφασίσατε να έχουμε στο κείμενο και το εξή. Υπενθυμίζοντα το ψήφισμα Β70531 του 2011 που κατετέθη βάσει του άρθρου 120 από την κυρία Μουσκαρδίνη και άλλους βουλευτές και εγώ έπρεπε να το πω αυτό, τώρα το έχω πει. Και για την τροπολογία 63 για τον φορολογικό, δημοσιονομικό φεδεραλισμό. Το κείμενο θα πρέπει να λέει θα μπορούσε να είναι χρήσιμο εργαλείο για να έχει μεγαλύτερη υποστήριξη. Είναι στη σελίδα 6 στο δικό μου κατάλογο ψηφοφορίας και μετά για να παρακολουθήσω αυτά που είπε ο το πρωί για τη συμβαστική τροπολογία 1α, αιτιολογική σκέψη ΤΣΙ, λατινικό, στη σελίδα 22 στο δικό μου κατάλογο ψηφοφορίας. Δεδομένου ότι το υπερβολικό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος πρέπει να λέει ε, έχει υποκαλέσει την κρίση. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές που έχω επιφέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μπλέξουμε όταν φτάσουμε στα σημεία αυτά θα μας υπενθυμίσετε τις αλλαγές όλε. Ξεκινάμε λοιπόν συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 3α υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 σε δύο τμήματα χωρίς τις λέξεις καταρχήν περιφερειακή αρρωγή, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Οι λέξεις περιφερειακή αρρωγή, υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά μήπως μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεύτερο τμήμα τη συμβαστική 4. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Γρήγορα, γρήγορα στο ψηφίσανε. Τώρα ένας από το ΕΛΚ περισσεύει. Ένας πρέπει να αποσύρθει από το ΕΛΚ, εντάξει, πέρας ψηφοφορίας και πράγματι απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 σε τμήματα, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, χωρίς τις λέξεις με ενδεχόμενη φορολογική εναρμόνιση, ψήφι υπέρ, το πρώτο τμήμα, κατά, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα, με τις λέξει και ενδεχομένω κάποια εναρμόνιση στα φορολογικά, υπέρ, κατά, αποχές. Και αυτό εγκρίνεται. 39, τροπολογία 39, υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Ένας από το ΕΛΚ περισσεύει και πάλι. Ευχαριστώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 2021. Προπολογία 38, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αφαιρέσαν την κάρτα από το ΕΛΚ. Ναι, μα το κάνανε. Ε, μ' αρέσει να ελέγχω, λέει η Αρλίν, για να είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι εντάξει. Αλλήν, σίγουρα δεν κλείνω ποτέ ψηφοφορία με μία κάρτα να περισσεύει. Αν τα ηλεκτρονικά δουλεύουν καλά και τα ηλεκτρόνια δεν πηγαίνουν όπου θέλουν, όλα πήγαν καλά. Τροπολογία 37 ψήφι υπέρ. Κατά. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 έλεγχος στη 42 άρχεται ψήφισατε όλοι πέρας με ισοψηφία απορρίπτεται 22-22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 κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 με προφορική τροποποίηση που ανέφερε ο Όλε Σμιτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 66 κάποια χέρια δεν σηκώνονται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβαστική 6α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά <clears throat> αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 ψήφι υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 84 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίθηκε. 23-21. 85 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε την 91 παρακαλώ Άρχεται η ψηφοφορία τώρα. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίψατε. 21 με 23. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κα, κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ Συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο στην παράγραφο 7. Ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 με προφορικό τμήμα που προστίθεται. Καταρχήν χωρίς την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροποποίηση ψήφι υπέρ. Την έχετε την τροπολογία. Είναι η τροπολογία των σοσιαλιστών λοιπόν υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η Ευρωπαϊκή Κομισιόν πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν στατιστικές για την φοροδιαφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι που υποστηρίζουν αυτή την τροπολογία υπέρ. Ο κύριος Ελχαντραούι, στην πραγματικότητα αυτή η προφορική τροπολογία επρόκειτο να συμπεριληφθεί ως προσθήκη στην συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 8 Νομίζω ότι είχε ψηφιστεί στη Συμβαστική 8 ήδη. Έτσι λέει ο κατάλογος της ψηφοφορίας. Εντάξει, πάντως συμφωνούμε για το κείμενο αυτό που θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Αν θέλουμε να το βάλουμε και στη σωστή παράγραφο. Και πράγματι νόμιζα ότι ήταν η παράγραφος 8. Μα ψηφίσουμε για την παράγραφο 8. Α, εντάξει. Ε, εντάξει. Αν δείτε τον κατάλογο, το είχαμε βάλει στη συμβαστική 8 Αλλά τώρα ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 9 η οποία αφορά την παράγραφο 8. Αν είναι σε λάθο θέση θα το μετακινήσουμε αυτό το κομμάτι. Ψηφίζουμε όμω, συμφωνούμε με αυτό, υπέρ, κατά, απόχε. εντάξει, το έχουμε δεχθεί και θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Είτε στο 8, είτε στο 9, είτε σε οτιδήποτε. 103. Τροπολογία 109. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά δεν κατάλαβα απόλυτα το έλθει την υποστηρίζει. Εντάξει, τότε περνάει. Πράγματος 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πράγματος 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 108 υπέρ στην παράγραφο 13, τροπολογία 108, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές 112, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 Παράγραφος μάλλον 16 υπέρ κατά, αποχές δεκτή, 113 υπέρ κατά, αποχές έλεγχος για την 113 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή για περιμένετε καταπίπτει καταπίπτει 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παράγραφος 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123, 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές καλύτερα να γίνει έλεγχος για την 127 ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας κατα... απορρίπτεται με 22-22 Αρχικό κείμενο παράγραφος 23 υπέρ κατά. Να ξαναδοκιμάσουμε. Παράγραφος 23 αρχικό κείμενο υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 134 ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 25 ψήφοι κατά 19 υπέρ 135 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά καλύτερα να ελέγξουμε έλεγχος για την 135 ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται 17 υπέρ 27 κατά 136 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά σας γίνει έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται 22-21 δίκαιο είχα που ελέγξαμε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται έλεγχος όμως για την 139 μήπως νομίζω ότι εγκρίνεται όμως 139 ηλεκτρονικός έλεγχος 139 Ψήφισαν όλοι, πέρας, απορρίπτεται. 20 υπέρ, 23 ψήφοι κατά. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δεκαβήτα σε δύο τμήματα. Χωρίς το αυτόματο. Πρώτο τμήμα χωρίς τη λέξη. Αυτή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά με τη λέξη αυτόματα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 150 σας παρακαλώ Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 27 κατά, 17 υπέρ. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα αν θέλετε. Απορρίπτεται. Κάπως λάθος μηνύματα πέρασαν πριν. Το δεύτερο τμήμα τη 153 απορρίπτεται λοιπόν. 154 υπέρ. Υπέρ τη 154. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Νομίζω ότι μόνο το έλκυνε κατά. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Ψήφισαν όλοι. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Πέρας. Εγκρίνεται 26 με 18. συμβεβαστικη 11 11α σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 δι λατινικό σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές υπέρ, νομίζω ότι εγκρίνεται. Η 164 εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά αποχές δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά να γίνει έλεγχος για την 166. Ψηφίσατε όλοι πέρας 21 ψήφοι υπέρ, 23 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος σας γίνει για την 169. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 26 ψήφοι υπέρ, 18 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται 170 υπέρ, κατά σύγχυσης. 170 υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 21 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καλώς. Ηλεκτρονικά ας κάνουμε την ψηφοφορία του τελικού κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 37 υπέρ, 5 κατά και μια αποχή. Ευχαριστώ λοιπόν. Συγχαρητήρια. Τώρα μόνο η προφορική ερώτηση που πηγαίνουν με τα, Euro, με τα ευρωμόλογα. Προφορική ερώτηση on block. Υπέρ. Ηλεκτρονικά θέλετε, καλώς. Άρχεται η ισοφορία. Οι απλές προφορικές ερωτήσεις που συνοδεύουν την έκθεση. Η ερώτηση, όχι το ψήφισμα. Εψήφισαν άπαντες πέρας. 42 υπέρ. Right, this might get complicated. Τώρα θα είναι κάπως πιο μπερδεμένο. Ψηφίζουμε για το σχέδιο ψηφίσματος. Ούντο. Πολύ ενδιαφέρον η μουσική. Ωραίος ο ήχος του κινητού. Συνάδελφοι, ευχαριστώ τον φίλο που μας επέτρεψε να μην είμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας και επιστρέψαμε σε κανονικές συνθήκες. Εδώ να πω ότι οι σκεώδεις εισηγητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους και προσπαθήσαμε να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση για τα ευρωομόλογα ώστε να συζητηθούν κατά έναν τρόπο αρμόζοντα από το Κοινοβούλιο. Σε αρκετές περιστάσεις η ομάδα μας επεσήμανε ότι δεν έχει υπάρξει ικανοποιητική η προσέγγιση, όπως τις συμβαστικές H, C και I, που λέγεται ότι είναι τόσο περίπλοκη διατύπωση, όπου δεν καταλαβαίνει κανείς τι θέλουμε να πούμε. Γι' αυτό λοιπόν δοκιμάσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα και προτείναμε κάποιες κατακμήματα ψηφοφορίες για να γίνουν λίγο σαφέστερα. Γι' αυτό λοιπόν, μισό λεπτό, μην πυροβολείτε, ε, σημειώνω ότι σε αντίθεση με μας Η παροχή των πληροφοριών δεν ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Δεν έλαβαν όλοι λοιπόν τις πληροφορίες εγκαίρως. Για να είμαστε σαφείς, στις συμβαστικές H, C και I. Τις αποσύρουμε τις τροπολογίες αυτές, τα απόσχουμε τις παραγράφους αυτές, μόνο και μόνο για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία. Και μετά ελπίζουμε ότι το κείμενο θα βελτιωθεί στην Ολομέλεια. Σιλβί. Ε, Πρόεδρε, για σκοπούς συμβιβασμού συμφωνούμε απολύτω να γίνει αυτό που προτείνει ο συνάδελφο, αλλά προσωπικώ αυτό που είναι σημαντικό για μένα και ευχαριστώ και τον Έντουαρτ Κλούνα και όλου του υπόλοιπου Κιώδη, είναι να δώσουμε ένα μήνυμα εγκαίρω στην Επιτροπή. Ένα μήνυμα κοινό από το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν να προχωρήσουμε άμεσα στι ψηφοφορίε. Ευχαριστώ. Αυτό που είπες είναι ότι δεν στηρίζεις τις συμβαστικές H, C, και I. Σωστά. Αλλά θες και κατά τμήμα ψηφοφορίες. Όχι, τις στηρίζουν χωρίς να τις ψηφίζουν. Δεν μπορεί τώρα να εμποδίζει τον ομιλητή <clears throat> πρόεδρος. Θέλαμε το H, το C και το 1 να τα κάνουμε σε χωριστή ψηφοφορία. Τώρα τα αποσύρουμε γιατί θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι δεν είχαν δυνατότητα στην ομάδα εργασία να τα συζητήσουν εγκαίρω και αυτή τη φορά δεν θα ζητήσουμε χωριστή ψηφοφορία και θα κρατήσουμε στάση αποχή. Είναι σαφέ αυτό ή πρέπει να το πω σε μια άλλη γλώσσα. Εντάξει. Τώρα κατάλαβα. έμπλεξα λίγο τις τροπολογίες με τις κατατμήματα ψηφοφορίες. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική C1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. E. Ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. I, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. K, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νάτι. L, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογικές ε, σκέψεις A, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη A, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική B, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της, ε, του ψηφίσματος. Υπέρ, Μάλλον ψήφισαν πάντες 37 υπέρ, 3 κατά, 4 εποχές. So now we move on. Πάμε τώρα. I can't see you. Να προχωρήσουμε. For the votes, they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 Are we, are we ready? Έτοιμοι. Λοιπόν, ξεκινάμε ψηφοφορία για το πλαίσιο εταιρική διακυβέρνηση για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Συμβαστική A, α, υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. think what you do is you. Right, do I, I, I, I, I, I the first I'm part. not sure whether everybody knows there's an oral amendment I think here. They do, the groups do. Okay, so we've now. could, could, could, could members listen, please? Μπορείτε να μ' ακούσετε. Τροπολογία 5 σε δύο τμήματα. Και υπάρχει και προφορική τροπολογία για το δεύτερο. Εκεί γίνεται την προσθήκη όπου δει πριν τους άλλους ενδιαφερομένους. Πρώτο τμήμα. Το δεύτερο λέει για τους εργαζομένους, τους μετόχους και όπου δει για τους άλλους ενδιαφερομένους. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επτά υπέρ, κατά αποχέ, απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική B υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Όχι, ωραία. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 γιατί δεν καταλαβαίνω κάτι είναι σκιασμένη. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω να διαβάζω. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα Συμβαστική D υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο, ε, συγγνώμη, τροπολογία 30 υπέρ. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. πάλι το όπου δει. Η ίδια τροπολογία με την προηγούμενη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κάτι έχει διαγραφεί εδώ, οπότε πάμε στην 36. 36. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 6 όχι, κάτι άλλο. Εγκρίθηκε, οπότε καταπληκτή. 39 υπέρ. Δύο τμήματα εδώ. Με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44. Με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική ε, ή υπέρ κατά αποχές. Πενήντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 51 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 52 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τελική εκδοχή. Εψήφισαν άπαντες πέρα της ψηφοφορίας. 26 υπέρ 12. 5 μάλλον κατά, 12 αποχέ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ωραία. Να θυμίσω σε όλους ότι μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής υπάρχει κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων από τις 6.30 έως τις 8 στο 6Q2. 6Q2 στο κτίριο Γιάν. Και τώρα παραδίδω την Προεδρία στον Θείοντορ. Συνάδελφοι, όσοι θέλουν να φύγουν παρακαλώ να φύγουν. Έχουμε και άλλες δουλειές σήμερα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Ελένα Μπασέσκου για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης των Λογαριασμών. Δίνω το λόγο στην κυρία Ελένα Μπασέσκου να παρουσιάσει το σχέδιο νομοδότησής της. Σιωπή παρακαλώ ησυχία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός ο... αυτή η πρόταση κανονισμού έχει ένα πολύπλοκο αντικείμενο, θέλει να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή διαδικασία για τον μπλοκάρισμα των λογαριασμών. <clears throat> Αυτό είναι εναλλακτικό για την εθνική διαδικασία, θα επιτρέψει να εμποδιστεί η απόσυρση καταθέσεων ή μεταφορά ε, ενεργητικών από οποιαδήποτε τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή η εσωτερική αγορά δίνει τη δυνατότητα μεταφορής ε, ποσών από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα σχεδόν ακαρία. Και με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να αποφύγει την πληρωμή <clears throat> χρεών. Αλλά δεν μπορούν οι πιστωτές να μπλοκάρουν με την ίδια ταχύτητα τους λογαριασμούς ενός ε, οφειλέτη τους στο εξωτερικό. Μπορεί να έχουν επίσης δυσκολία να κατανοήσουν πού βρίσκεται ο λογαριασμός του οφειλέτη αν βρίσκεται σε μια άλλη χώρα. Ο κανονισμός αυτός θα επιτρέψει να εμποδιστούν οι μεταφορές πιστώσεων ή οι αποσύρσεις κονδυλίων από οποιοδήποτε τέτοιο λογαριασμό και θα εφαρμόζεται και στις διαδικασίες που είναι σε δικαστική διαδικασία ή και αυτές οι οποίες είναι σε διατησία. Έχουν παρουσιαστεί 27 τροπολογίες από εμένα ως εισηγήτρια. Νομίζω ότι φέρνουν καλύτερη διαφάνεια σε ορισμένες πρόνοιες του σχεδίου κανονισμού και από οικονομική και από νομική πλευρά. Ο κύριος στόχος μου να εξασφαλίσω μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των οφειλετών και την προστασία που πρέπει να τύχουν και των δικαιωμάτων των ε, πιστωτών για να ανακτήσουν μένα ποσά και έτσι να μειωθούν οι δυνατές καταχρήσεις. Προτείνω με την τροπολογία 1 να υπάρξει και κάποιο ποσό ασφαλείας, κάποια εγγύηση η οποία θα καθορίζεται από το αντίστοιχο δικαστήριο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξουν κάποια κριτήρια για να αποφασίζεται το επίπεδο των απαιτήσεων εναντίον ενό οφειλέτη. Η τροπολογία 3 δίνει εξαιρέσει από το, τη σφαίρα εφαρμογής για να υπάρξει η λειτουργία του συστήματος και υπάρχει απλώς ένα σύστημα για το συμψηφισμό των εγγύησεων. Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε συνέχεια στις ε, διατάξεις οδηγίας 91-426. Θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της ταχύτητος που αναφέρεται σε πολλές τροπολογίες οι οποίες προτείνουν μια σειρά από καταληκτικές προθεσμίες προτείνω να αναφέρονται ημερολογιακές ημέρες στις τροπολογίες 15, 19 και 25. Στην τροπολογία 20 προτείνω επίσης ο φιλέτης να του κοινοποιείται μέσα σε μία εργάσιμη μέρα το γεγονός ότι υπάρχει μια εντολή κλεισίματος του λογαριασμού. Και επίσης θέλω να διευκρινίσω πότε υπάρχει διαμεθοριακός χαρακτήρας μιας υπόθεσης. Και να είναι σαφές πότε οι υποθέσεις μπορεί να έχουν διαμεθοριακό, διαμεθοριακή πτυχή η τροπολογία 21 καθώς και η τροπολογία 22 τροποποιούν το άρθρο 26 που αναφέρεται <clears throat> στην ε, απόφαση για την εντολή μπλοκαρίσματος και η παράγραφος 4 του αρχικού κειμένου δεν ήταν επαρκώς σαφής σε σχέση με τις ισοτιμίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση που τα χρήματα βρίσκονται σε διαφορετικό νόμισμα από τον νόμισμα της χώρας στην οποία εκδόθηκε η διαταγή μπλοκαρίσματος του λογαριασμού. Στην τροπολογία 26 προτείνω η μετατροπή των νομισμάτων να γίνει από την ίδια την τράπεζα όπου είναι τα χρήματα και αυτό βάσει το τιμία της κεντρικής τράπεζας στις τοποθεσίες της χώρας όπου βρίσκεται αυτή η τράπεζα. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί αλλιώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη τιμή αναφορά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που βασίζεται στον μέσο όρο των συναλλαγών τη Κεντρική Τράπεζα. Η τροπολογία 21 στο άρθρο 26 διευκρινίστε καλύτερα η κατάσταση τι γίνεται αν ξεπερνάνε τα ποσά σε ένα λογαριασμό το ποσό το οποίο αναφέρεται στην ε, εντολή μπλοκαρισμού του λογαριασμού, τότε η τράπεζα θα πρέπει να αποφασίσει σε ποια στοιχεία του ενεργητικού εφαρμόζεται η εντολή αυτή μπλοκαρισμού. Στο τέλος να σας δώσω μερικές πρακτικές ε, λεπτομέρειες. Στις 12 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα συζητηθούν στην συνεδρίασή μας στις 6 Φεβρουαρίου. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 28 Φεβρουαρίου. Περιμένω λοιπόν για τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας και είμαι διαθέσιμη για να τις συζητήσω. Ο κύριος Μπούλμανος και ο δισηγητής έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και σας κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα σημαντικό μέτρο για την εσωτερική αγορά, ένα σημαντικό νομικό μέτρο. Δεν θέλουμε να επιτρέπουμε αυτοί που έχουν νόμιμες απαιτήσει να μην μπορούν να τις εφαρμόσουν λόγω της διαφοράς ε, από τη μία χώρα στην άλλη των διατάξεων που ισχύουν για το μπλοκάρισμα του, των λογαριασμών. Θέλουμε λοιπόν με αυτόν τον επικοδημητικό τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτή την πρόταση και υποστηρίζουμε αυτά τα οποία λέει και η προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζουμε ότι θα είναι σημαντικό αυτό το οποίο θα αποφασίσουμε για να εξασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία. Από τη μία την πλευρά μεταξύ των αναγκών αυτών που έχουν μια απέτηση επί των οφειλετών και επίσης την προστασία ενός ε, λογαριασμού ο οποίος θα βαρύνεται με μια εντολή αποκλεισμού και αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα σε καταναλωτές, σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν πρέπει να μείνουν χωρίς ένδικα, χωρίς νομικά μέσα για να μπορέσουν να αντισταθούν σε μια τέτοια εντολή και οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να προσφύγουν στη δική τους εθνική τάξη. Δεν θέλουμε όμως συγχρόνως να υπάρξει απόκρυψη και συσκότηση για τα θέματα αυτά και να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο κλείσιμο το λογαριασμό χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς γίνεται. Θα πρέπει η νομική λοιπόν οργάνωση να είναι τέτοια ώστε και οι δύο πλευρές να έχουν την κατάλληλη ισορροπία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Θα διατυπώσουμε τροπολογίες που θέλουμε να είναι απόλυτα θετικές προς την κατεύθυνση που υπέδειξε η εισηγήτρια ώστε να μπορέσει να τεθεί το ταχύτερο δυνατό σε εφαρμογή αυτό το νομικό μέτρο. Κάποιος θέλει να αντικαταστήσει την κυρία Γκουλάρ η οποία είναι απούσα. Όχι. Ο κύριος Στρίτσεκ. Ούτε και αυτός είναι πάρα. Κύριε Γκίκολτ, έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε για την έκθεση. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα ήδη υπόθηκαν. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο συστατικό αυτό και ένα χρήσιμο συστατικό προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά. Επίσης θεωρούμε ότι η έκθεση είναι καλή. Στηρίζουμε τη γενική της κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ασφάλειας και θα πρέπει να υπάρξει κάποια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Σε γενικές όμως γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι με την έκθεση. Ευχαριστούμε. Ο Τόμα Χέντελ. Δεν είναι εδώ. Κάποιο άλλο που θέλει το λόγο εκ μέρου του. Okay, Κύριε Γκοζέ, κύριε Πρόεδρε, απλώ να πω το εξή προς την εισηγήτρια που έχει κάνει εξαιρετικό έργο ότι η ομάδα του ΕΛΚ θα τα στηρίξει. Thank Σας ευχαριστούμε. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Κυρία Μπασέσκου, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Πολύ ωραία. Δεν θέλει. Κλείνουμε το σημείο αυτό. 12 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι, τροπολογίες. Σχέδιο έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων της έκθεση 2010 από τον κύριο Καμάλ. Κύριε Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Ε, ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, μια από τις αρχές της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών είναι να φροντίζουμε να μην πηγαίνει χαμένο το χρήμα των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό βλέπω και να χαμογελάνε οι συνάδελφοι στην αίθουσα. Βεβαίω και με τη διαφάνεια τα πάμε καλά, όπω και οι πράσινοι. Είναι ένα από τα πράγματα με τα, για τα οποία συμφωνούμε με τον Πασκάλ. Εδώ βέβαια θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε κάποια στοιχεία, αλλά τα έχουμε σχεδόν καταφέρει. Ξεκινώ με την εξή αρχή. Ότι θα πρέπει ότι οι πολίτε των ευρωπαϊκών χωρών να γνωρίζουν πώ δαπανώνται τα χρήματά του και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια η σύγκληση των δημοσιονομικών διαπαιτήσεων θα μεταβληθούν λόγω της συμφωνίας μεταξύ κατών μελών και θα επηρεαστούν και κεφαλαιοκές αγορές παγκοσμίω. Οι, δια... διαθετήσεις αυτές βεβαίως θα πρέπει να είναι αδιάβλητες. Το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε την έγκρισή του για τον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και τη λειτουργία της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. πάντω, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η λειτουργία της τράπεζας αυτής είναι και σε συντονισμό με την ε, στρατηγική του 2020 και δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη, επανάληψη των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε και την έκθεση στον κίνδυνο, καθώς και τα προγράμματα που θα καλύπτονται από την τράπεζα αυτή και θα πρέπει να συμβάζεται και με τι διεθνεί προδιαγραφέ η τράπεζα, καθώ και να γίνει μια δοκιμή κοπόσεω, ώστε να βεβαιωθούμε ότι είναι ανθεκτική. Επίση, για τι μακροπρόθεσμε επενδύσει τη τράπεζα αυτή, θα πρέπει να δημοσιεύονται σε έναν ιστότοπο και να είναι σαφή στη θέση τη ω προ τα βασικά δημοσιονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την κατάσταση υγεία τη Ευρωζώνη. Ένα ζήτημα περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα που θα πρέπει να επικεντρώσει τι προσπάθειέ τη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ξέρω βέβαια ότι εδώ έχουμε απλώ ένα σχέδιο έκθεση και ευχαρίστω να δεχτώ προτάσει. Είναι κατά πόσο θα πρέπει να στρέψει την προσοχή τη στι αναδυόμενε δημοκρατίε γύρω από τη Μεσόγειο, από την αραβική πλευρά τη θάλασσα αυτή. Ξέρουμε ότι η πραγματική οικονομία έχει δεχτεί σοβαρέ πιέσει λόγω των τριγμών του τραπεζικού τομέα, όμω θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει την μπορεί για να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο. Ελπίζουμε να είναι σταθερή και υπάρχουν εδώ και εκθέσεις από τα κρατημέλη. Υπάρχει έκθεση των κατομελών προς την τράπεζα αυτή. Ελπίζω ότι αυτές οι βασικές αρχές θα βρουν σύμφωνο στους περισσότερους συναδέλφους από όλες τις ομάδες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καμάλ. Ένα είναι ο Σκιώδης. Εισηγητής η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Καμάλ για τις ε, παρατηρήσεις του και για τα θέματα που έχει θίξει. Συμφωνώ με όλους ε, τους στόχους που θέτει, την καλύτερη αξιοποίηση ε, των χρημάτων της Ευρωπαϊκής, κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και συμφωνώ με τα, αυτά που ήδη το σχέδιο γνωμοδότησης μας επισημαίνει, καταρχάς την αποτελεσματικότητα και το συντονισμό με τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τα διαρθρωτικά ταμεία θα σημειώσω ιδιαίτερα για την επίτευξη των στόχων ε, όσο και για την ε, διατήρηση της αξιολόγησης ΑΑΑ. Το έχουμε τόσο ανάγκη τον τελευταίο καιρό να το επισημαίνουμε αυτό το, το 3α. Ε, και από την άλλη πλευρά ε, συμφωνώ και με την εξωστρέφεια της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως τονίστηκε κυρίως στην νότια ακτή. Αυτά που ήθελα να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι έχουμε ανάγκη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προάγει την ε, καινοτομία ιδιαίτερα, θα το τονίσω αυτό με τροπολογίες, ε, την καινοτομία όπως ήδη αποτελεί από το 2000 στόχους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και επενδύει κεφάλαια στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και την εφαρμογή της στην αγορά. Θα το τονίσω αυτό. Επίσης θα τονίσω ιδιαίτερα ε, την, ε, τα προγράμματα, το Jeremy και το Jasper στο πρόγραμμα ε, και το, το Jasmine, το Jessica επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά διότι δίνουν την ευκαιρία στην μεγιστοποίηση των πόρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την πολιτική συνοχής και την ε, διευκόλυνση των κρατών μελών, κυρίως των χωρών με τις δημοσιονομικές δυσκολίες σήμερα, για να συντονίσουν τις χρηματοπιστωτικές τους ανάγκες και δυνατότητες προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Ε, έχω να τονίσω αυτό ιδιαίτερα και επίσης ε, ως προς την επέκταση για την νότια ακτή θέλω να χαιρετήσω διότι αναφέρει την ανάγκη ε, ο κύριος Καμάλ ε, να φέρει καλή την τράπεζα να εντείνει τις δραστηριότητε της. Πρέπει να τονίσουμε ότι έχει μια μακρά πείρα με το ΦΕΜΙΠ, ένα ειδικό όργανο ε, για την ευρωμεσογειακή συνεργασία η τράπεζα. Έχει ήδη ενισχύσει με ένα δισευρώ στο πλαίσιο του Arab String τα κεφάλαια που διαθέτει και επίσης συμφωνώ με ε, το συντονισμό, το αναφέρει ο κύριος Καμάλ νομίζω, το συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η οποία ήδη δραστηριοποιείται στην νότια, στην όχθη της Μεσογείου. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα θέματα που θέλω ή να επισημάνω ή να συμπληρώσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, σας ευχαριστώ καταρχάς. Υπάρχουν και άλλοι ε, σκιώδεις εισηγητές και θα ήθελα ε, να τακτοποιηθούν κάπω τα ονόματα. Δεν έχω μπροστά μου τα ονόματα. Ο κ. Κούτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καμάλ για το κείμενό του, για τη γνωμοδότηση και θα ήθελα να του πω ότι και η δική μου ομάδα μάχεται για να δώσει υπεραξία στα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. χρειάζεται ένωση οικονομική ανάπτυξη βάσει έρευνας, εκπαίδευσης, μεγάλων επενδύσεων, καινοτομίας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να αποτελέσει έναν παράγοντα και ένα εργαλείο για να βγούμε από την οικονομική αυτή κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό αυτά τα διάφορα, τα project bonds όπως αποκαλούνται, ε, έχουν σαν στόχο τη συμπληρωματική χρηματοδότηση και θα πρέπει να λειτουργήσουν το ταχύτερο δυνατόν ή δυνατόν πριν από την περίοδο 2014-2020. Θα ήθελα να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου για την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την παροχή τεχνικής βοηθείας προς τα κράτη-μέλη εκείνα που έχουν πρόβλημα ε, όσον αφορά την χρήση και απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων είναι πολύ καλή ιδέα και μπορεί να υποστηρίξει έτσι περαιτέρω τις χώρες, τις προσπάθειες που καταβάλουν για να αναπτυχθούν. Και κάτι άλλο με το οποίο συμφωνώ ε, όσον αφορά αυτά που είπε ο αφορά την πολιτική διαφανείας ε, της τράπεζας. Είναι πρόσδεκτο ότι το 2010 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υιοθέτησε ένα νέο πλαίσιο αρχών και πρακτικών όσον αφορά τη διαφάνεια. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τις εκθέσεις περιβαλλοντικών ε, επιπτώσεων ε, και να δημοσιεύονται πριν εγκριθούν οι εκθέσεις αξιολόγησης συνεπιών. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και επί της ανάγκης που υπάρχει η τράπεζα να διενεργεί ανεξάρτητη αξιολόγηση των νομολογιών των οποίων δραστηριοποιείται για να αποφευθούν οι παράνομες οικονομικές ροές και η οικονομική παράδειση. Προσβλέπω στη συνεργασία με τον κύριο Καμάλ και με τους άλλους συναδέλφους επί του ζητήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κούτας. Ο κύριος Κυλακάκης έχει το λόγο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα λέω ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πολύ καλό περιεχόμενο της έκθεσής ε, του. Θέλω να προσθέσω μερικά ακόμα στοιχεία για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θέτων έμφαση στις χώρες που καλύπτονται από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και παίρνουν υποστήριξη <laughs> από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει αλλάξει το παιχνίδι για τις χώρες αυτές. Μιλάμε για μια τελείως διαφορετική οικονομική κατάσταση και το κύριο, το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές είναι να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την εισρωή επενδύσεων και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος εταίρος για επενδύσεις για τις χώρες αυτές, γιατί με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για να επιτύχουν τα προγράμματα αυτά. Και αυτό πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό γιατί οι νέες επενδύσεις στις χώρες αυτές, όπου υπάρχουν τεράστια προβλήματα ανεργίας, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες ούτως ή άλλως και θα αποτελέσουν και ένα μήνυμα ότι τα προγράμματα αυτά προχωρούν επιτυχώς και προς την επόμενη φάση τους. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, και αυτό είναι κάπως πιο μακροχρόνιο, είναι ότι τώρα που θέλουμε να δημιουργήσουμε μια δημοσιονομική ένωση, η οποία θα έχει μεγαλύτερο χαρακτήρα αφαιστηρότητος σε σχέση με τα ε, μέσα και τα εργαλεία που θα έχουν τα κράτη, μέλη και οι κυβερνήσεις τους, Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να παίξει και κάποιο ρόλο μεγαλύτερο σε χώρες ή σε περιοχές οι οποίες έχουν εμπλακεί σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής επένδυσης, χαμηλής παραγωγικότητας, χαμηλής καινοτομίας. Γιατί οι χώρες, οι, οι περιοχές που βρίσκονται σε δημοσιονομική στενότητα και δυσκολία δεν έχουν και τόσα πολλά εργαλεία στην φαρέτρα τους για να μπορέσουν βέλη βέλτιστη φαρέτρωση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά και όταν έχουμε ένα ασυμμετρικό κλειδονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετικά τα αποτελέσματά του στι χώρε του κέντρου και στι χώρε τη περιφέρεια. όπου η οικονομία των περιχώρων αυτό δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και γι' αυτό χρειαζόμαστε να έχουμε τα εργαλεία που θα βοηθήσουν την περιφέρεια να εξέλθει από την κρίση και το σοκ. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να παρατηρεί να συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τροποποιήσει τις σκέψεις γιατί μακροπρόθεσμα θα χρειαστεί να έχουμε τον τρόπο να βοηθήσουμε τις περιφέρειες και τις χώρες αυτές να προωθήσουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα ελήψη άλλων εργαλείων στη διάθεσή τους. Με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευχαριστώ. Πρωτού δώσω το λόγο στην, στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα ήθελα να ξέρω αν κάποιο άλλο δεν θέλει να λάβει το λόγο. Ο Πασκάλ. Σας σκιώδης για τους πρασίνους θα μιλήσω. Η ομάδα των πρασίνων ε, υποστηρίζει πολύ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μονίμως προσπαθούμε να δώσουμε τα καλύτερα μέσα στην τράπεζα αυτή για να κινείται. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε λοιπόν ε, ποια είναι η θέση της όσον αφορά το σεβασμό της Βασιλείας 3 κατά πόσο στα κείμενα που όπως έχουν συνταχθεί σήμερα αν περιέχονται κάποια στοιχεία που δημιουργούν προβλήματα για μια τράπεζα που έχει ειδικές, ε, ειδική αποστολή και ειδικό σκοπό. Ε, οπότε στις τροπολογίες θα θέσουμε ερωτηματικά σε αυτά που προτείνει ο εισηγητής ο Καμάλ, ότι θα πρέπει υποχρεωτικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, θα πρέπει να, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις στο μέλλον. Θα θέλαμε και ποια είναι η άποψη τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επ' αυτού. Ε, δεύτερον, όσον αφορά το κεφάλαιο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, Επενδύσεων, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, αντίθετε εξελίξει σε αυτή τη φάση. Έγινε μια αύξηση μετά την κρίση και μετά ακολουθείται διαφορετική κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μαζί να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ενισχυθεί οικονομικά για να μπορεί να δράσει κατά τη υφέσεω, αλλά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και επί επενδύσεων που θα συνάδουν με τους στόχους που έχουν καθοριστεί από τις συνθήκες και κυρίως τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσης του 2020 που υπενθυμίζει ο εισηγητής. Ίσως τελευταίο σχόλιο που ίσως θα δικαιολογούσε κάποιες τροπολογίες σχετικά με την ενεργειακή πολιτική είναι μια συζήτηση που διεξάγεται μονίμως με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα θέλαμε το έγγραφο που καθορίζει τους πολιτικούς ενεργειακούς ε, προσανατολισμούς να ταιριάζει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσης, κυρίως τους στόχους για το κλίμα που έχουν καθοριστεί για το έτος 2050, που αυτό ίσως να συνεπάγεται επιλογές επενδυτικές και χρηματοδοτικές διαφορετικές από αυτές που γίνονται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος Ευρωβουλευτής. Θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Κουζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να θέσω ένα ερώτημα. Τη θέτω προς την εισηγητή για να διερωτηθεί και αν είναι πρόσωπος Ευρωπαϊκής Τράπεζας απαντήσει καλό. Και εδώ συμπληρώνω κάπως το ερώτημα του Πασκάλ όσον αφορά τι δυνατότητε που έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από ό,τι γνωρίζει το κεφάλαιο τη δεν είναι, έχει ελευθερωθεί πλήρω το κεφάλαιο τη ε, υπό τι παρούσε περιστάσει που έχει μετόχους ε, η τράπεζα αυτή που περνούν ε, δύσκολες οικονομικές καταστάσεις αν υπάρχει δυνατότητα να, να ε, μην εμποδίζεται η χρηματοδότησή της από αφιβολίες που ίσως υπάρχουν από τη δυνατότητα που έχουν οι μέτοχοι να σεβαστούν τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που υπάρχουν για την απελευθέρωση του κεφαλαίου των πόρων. Ευχαριστώ ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και θέλω ευχαριστώ και τον εισηγητή σας και τους σκιώδεις εισηγητέ και τους υπόλοιπους βουλευτές για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους, όλες τις από τις οποίες καταγράφουμε και φυσικά θα λάβουμε υπόψη για την περαιτέρω εξέλιξη των εργασιών μας. Για να σταθώ σε αυτά που είναι τα σημαντικά θέματα τα οποία γίνονται σήμερα. Η λογοδοσία. Νομίζω ότι γνωρίζετε πόσο ο πρόεδρος Μέισταρ κατά τη διάρκεια των 12 ετών του επικεφαλής της τραπεζάς μας έχει δώσει έμφαση στη λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την έποψη αυτή έχουμε αναπτύξει και ένα μνημόνιο κατανόησης σχέδιο μνημονίου, δηλαδή μεταξύ της τράπεζάς μας και του Κοινοβουλίου για να ε, διαρθώσουμε καλύτερα αυτή τη λογοδοσία και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί του χρόνου. Και ο πρόεδρος ε, Μέιστατ επίσης υποσχέθηκε χθε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να δώσει μέσα στην αρχή του 2012 μία έκθεση για την χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων μας και επομένως όλα στρέφονται προς την κατεύθυνση που αναφέρατε για τη διαφάνεια. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στη νέα πολιτική στην οποία έχουμε καταλήξει και η οποία έχει δημοσιευτεί μετά από μακρές διαβουλεύσεις και ελπίζουμε ότι θα ικανοποιήσει και την αίτηση της διαφάνειας. Παραμένουμε πάντα για περαιτέρω βελτιώσεις. Για θέματα πολιτικής νομίζω ότι θα ήταν ορθό να εστιάσουμε την προσοχή μας στην επίτευξη στρατηγικής Ευρώπη 2020, μια <clears throat> ευφυής βιώσιμη και περιεκτική μορφή ανάπτυξης. Εκεί πρέπει να δώσουμε όλους τους πόρους μας και την ικανότητά μας και αυτό το ενέκρινε το Διοικητικό μας Συμβούλιο πρόσφατα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Τραπέζας Επενδύσεων είναι δύσκολη καιρή, είναι πολύ πολύπλοκα τα πράγματα <clears throat> κατ' ουσίαν φυσικά λαμβάνουμε υπόψη πλήρως τι διατάξεις της Βασιλείας 3 στο βαθμό που εφαρμόζεται στις δραστηριότητές μας. Βέβαια δεν είμαστε εμπορική τράπεζα, δεν δίνουμε στεγαστικά δάνεια, δεν έχουμε καταθέσεις και καταναλωτικά δάνεια όπως μια εμπορική τράπεζα, αλλά σίγουρα λαμβάνουμε υπόψη την ουσία της Βασιλείας 3 και από την Επιτροπή μας που είναι υπεύθυνη για τους λογιστικούς ελέγχους. Θεωρούμε ως γνώμονα γιατί βρισκόμαστε μέσα στα πλαίσια των συνθηκών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνουμε σαν νομική βάση πάντα όλα αυτά που περιλαμβάνονται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως θα έχουμε και την οδηγία CRD το ταχύτερο δυνατό που θα την εφαρμόσουμε. Τι είναι αυτό το οποίο, στο οποίο οφείλεται το τριπλό α της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τρία πράγματα. Η ισχύς των μετόχων μας, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και η περιφερειακή κατανομή των στοιχείων ενεργητικού μας. Γνωρίζουν όλοι ότι είναι ισχυρή η μετοχή μας. Βέβαια έχουμε τα ίδια προβλήματα όπως οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, κοινών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά το χαρτοφυλάκιό μας μένει ισχυρό. Δεν υπέστημε καμία σοβαρή ζημιά και οι πιο δύσκολες περιπτώσεις που παρακολουθούμε προσεκτικά ουσιαστικά έχουν υποστεί ζημίες της τάξης του 1-2% μονάχα. Τώρα βέβαια, όταν η ποιότητα των μετόχων μας βρίσκεται υπό πτωτική πορεία, τότε οι εταιρείε αξιολόγησης κοιτούν περισσότερο τα βασικά, τον βασικό λόγο κεφαλαίων στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερο κεφάλαιο για να είμαστε επαρκή στα μάτια των αγορών. Εδώ χρειαζόμαστε νέα πνοή ζωή και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ή θα πρέπει να αυξήσουμε του κεφαλαιοχικού μα πόρου ή θα πρέπει να μειώσουμε τι δανειοδοτήσει μα. Δεν υπάρχει καμία ε, άλλη δυνατότητα. Υπάρχει αριθμητής και παρανομαστής και για να διατηρήσουμε το λόγο αυτό σταθερό θα πρέπει να κάνουμε ή το ένα ή το άλλο. Επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο Τη τράπεζα αποφάσισε να μειώσει τι δανειοδοτήσει που προβλέπεται να δώσουμε στα επόμενα τρία χρόνια, κάτι το οποίο φυσικά είναι λυπηρό λόγω του ρόλου που έχει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά είναι ο μόνο τρόπο να διατηρήσουμε την δανειοληπτική μα ικανότητα. Και αυτό με φέρνει στην σημασία του να δημιουργήσουμε από κοινού με τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτικά ε, εργαλεία, γιατί έτσι μπορούμε να αμοχλεύσουμε καλύτερα το κεφάλαιό μας και όπως λέει ο κύριος ε, το να ζητήσουμε τώρα να καταβάλουμε το εγγεγραμμένο κεφάλαιο οι μέτοχοί μας είναι κάπως δύσκολο σε αυτή τη χρονική στιγμή. Είναι απαραίτητο να παίξει μεγαλύτερο ρόλο η αξιοπιστία μας ε, σε ενέργειες όπως τα λεγόμενα project bonds, όπου υπάρχει ουσιαστικά μια μόχλευση κονδυλίων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας τονίσω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης θέτει αυτή τη στιγμή τα project bonds δίπλα στα ευρωομόλογα, αλλά είναι διαφορετικά τελείως. Τα project bonds εκδίδονται από ιδιωτικέ εταιρείε για να υποστηρίξουν τι επενδύσει στα ευρωομόλογα. Ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα ότι είναι τελείω διαφορετικό θέμα, επομένω δεν έχουν καμιά σχέση με την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για τη Μεσόγειο. Φυσικά αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μα, αλλά δεν θα σα εκπλήξει αν πω ότι τα αποτελέσματά μας εφέτος δεν φτάνουν το επίπεδο των προσδοκιών μας, γιατί η πολιτική κατάσταση της χώρας αποδέκτριας δεν μας επέτρεψε να έχουμε τους σωστούς συνομιλητές για να μπορέσουμε να θέσουμε σε κίνηση τα διάφορα εγχειρήματα και σχέδια και τις δανειοδοτήσεις που θα θέλαμε να κάνουμε. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αφορά όλα τα χρηματοδοτικά ε, μέσα και φορείς που λειτουργούν στην περιοχή αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα θελήσουμε να κάνουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε τη δέσμευση της Ντοβίλ να δανείσουμε μέχρι 6 δισεκατομμύρια στην περιοχή το 2013, αλλά αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο και πιο μεγάλη πρόκληση μέχρι ότου ομαλοποιηθεί η πολιτική κατάσταση. Οι χώρες προγράμματος όπως ανέφερε ο κύριος Σκυλακάκης, αυτό είναι Πολύ σημαντικό για μας, εμείς αποδίδουμε μεγάλες προσπάθειες για το θέμα αυτό. Συζητούμε με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Θεμάτων, συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συνδυάσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία και τους πόρους που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να εκταμιευθούν με τη δυνατότητα <clears throat> δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Παιδίσεων μορφή εγγύησεων και διαμοιρασμού κινδύνου που θα επιτρέψουν για τις χώρες να εφαρμόσουν τα διαρθρωτικά αυτά και η τράπεζά μας να κάνει μεγαλύτερες δανειοδοτήσεις. Είμαστε σίγουροι ότι με τη μοστήριξη των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου σας θα μπορέσουμε του χρόνου εν καιρό να εφαρμόσουμε και αυτή τη νέα προσέγγιση. Τέλος για τα ενεργειακά θέματα, ναι, σας έχουμε ακούσει την άποψή σας, παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά του, το στόχο του 2050 τα τελευταία αποτελέσματα που είχαμε είναι ότι 75% της δανειοδότησής μας για ενεργειακά projects είναι για ανανεώσιμες ενέργειες. Αυτό είναι ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα. Από τα υπόλοιπα 10% αφορούν ενεργειακά σχέδια ορυκτών καυσίμων που δυστυχώς είναι και αυτά τα οποία εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί η πτυχή της ενεργειακής ασφάλειας σε περιοχές που δεν υπάρχουν Εναλλακτικέ λύσει, Στη Γερμανία, χάρη, το πρόγραμμα απόσυρση από την πυρηνική ενέργεια οδήγησε σε μια κατάσταση, ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρω από πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμε ενέργειε, οπότε χρειάζεται να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα γεφύρωση. Κάποια ερωτήματα για να υπάρξει μια διευκρίνηση και για μένα και για του άλλου. Είπατε ότι τα project bonds εκδίδονται από ιδιωτικέ εταιρείε ποια είναι η σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των project bonds αυτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να το αποσαφηνίσω περαιτέρω. Το θεμελιώδες αυτό θέμα των project bond για την εξαγωγή ενέργειας ή σχέδια τηλεπικοινωνιακά. Αυτά πολλές φορές ε, εφαρμόζονται μέσω μια εταιρική σχέσης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, PPP όπως λέγεται. Εφόσον είναι το κατάλληλο μέσο για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή εφόσον μια εταιρεία θέλει να μαζέψει κονδύλια, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα project bonds. Δεν έχει όμως την πιστοτική αυτή ικανότητα ώστε να προσελκύσει τα τεράστια ποσά που μπορεί να Υπάρχουν από ασφαλιστικέ εταιρείε, από επενδυτικέ, από την αγορά. Εδώ λοιπόν μόνο με καλής αξιολόγηση υψηλή ποιότητας bonds, ομόλογα μπορεί να γίνει αυτή η συλλογή κονδυλίων. Είναι λοιπόν ένα δάνειο αυτό σε χαμηλότερο επίπεδο Οπότε ουσιαστικά τροφοδοτούμε πιστοτικά το ομόλογο και βελτιώνουμε την ποιότητά του. Οι θεσμικοί λοιπόν παράγοντες κάποια στιγμή ενδιαφέρονται και αγοράζουν. Με ένα λοιπόν δευτερογενές δάνειο, το οποίο μπορούμε να πάρουμε μόνο από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, έτσι καταφέρνουμε και βελτιώνουμε την ποιότητα των ομολόγων. Με 4-5 εκατομμύρια τον προπολογισμού χοντρικά μπορεί κανείς να αντλήσει 20 εκατομμύρια περίπου δευτερογενή δάνεια από την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων με δυνατότητα χρηματοδότησης 100 εκατομμυρίων που θα καλύψουν προγράμματα των 150. Αυτή είναι η δυνατότητα μόχλευσης που έχουμε. Η εταιρεία είναι ο φιλέτης μετά. Η ιδιωτική εταιρεία. Μάλιστα, να επανέλθω στον εισηγητή αν θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ τους Κιώδης και τους άλλους ε, και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις απόψεις που εκφράστηκαν. Θα λάβω υπόψη πολλά από αυτά που υπόθηκαν. Περιμένω τροπολογίες. Ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο που προφέρω τα ονόματα από την κυρία ε, Κράτσα. Την ευχαριστώ για αυτό που είπε για την Νότια Αχτή, για τη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι επί το οποίο διαφωνούμε. Γνωστοποιήστε το μου αν διαφωνούμε κάπου. Περιμένω τι τροπολογίε σα. Ε, ευχαριστώ πολύ ε, και Σούτας. Ε, πρέπει να έχουμε υπεραξία στα χρήματά μας. Περιμένω και δικές τροπολογίες. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν οι χώρες αυτές που έχουν ταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Μπορώ να μιλήσω μαζί σας. Ο κ. Σκάλφα, συνεργαζόμαστε ως συνήθως συζητάμε γιατί θα αμφισβητήσετε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να συμμορφωθεί με τη Βασιλεία 3. Ε, ίσως υπάρχει παρεξήγηση, μπορεί να το συζητήσουμε ε, το θέμα. Κατανοώ την ενθάρρυνση χρήσεως ανανεωσίμων πηγών ενεργείας. Αυτό που έθεσε ο κύριος Γκοζές ετέθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο από Βρετανό βουλευτή. Δηλαδή, τι άλλες ευθύνε έχουν τα κράτη-μέλη ε, όταν ζητείτε κεφάλαιο. Αυτούς δύσκολους καιρούς φαίνεται να μην είναι ρεαλιστικό το αναμενόμενο ποσό. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και τέλος, αυτά τα project bonds. Τι πρέπει να συζητήσουμε, αν όχι σε αυτό, ίσως σε άλλο πλαίσιο. Είναι ποιο πλήττεται πρώτος δεν είναι πάντα ο ιδιωτικό επενδυτή που πλήττεται, αλλά οι φορολογούμενοι που πληρώνουν πρώτοι και θα πρέπει πιστεύω να συμφωνήσουμε όλοι ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Περιμένω λοιπόν και τις τροπολογίες, συζητήσει και με τους Κιώδη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και α ξεκινήσει η μάχη λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καμάλ. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Εισηγητής ο κ. Κλούτερ. Του δίνω ευθύς αμέσω το λόγο. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει μείνει πολλοί κόσμος, παρόλα αυτά μπορούμε να συνεχίσουμε. Το θέμα της ε, χρηματοπιστωτικής περιεκτικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό η έκθεση αυτή έχει κατανεμηθεί πριν από ένα χρόνο περίπου μεταξύ των συντονιστών. Είχε καθυστερήσει κάπως η απόδοση αυτής της έκθεσης γιατί άλλαξε η Επιτροπή μας την άποψή της και αποφάσισε αντί για έκθεση να έχουμε μια σύσταση. Και μετά από αυτή την ε, σύσταση χρειάζεται ένας χρόνος ελέγχου εφόσον απευθύνεται στα κράτη-μέλη για να δούμε κατά πόσο μπορούν να εξασφαλίσουν την κατάλληλη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στις τραπεζικές υπηρεσίες. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η δυνατότητα ελέγχου για ένα χρόνο παρακολούθησης. Αποφασίσαμε ως συντονιστές ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε σε κάτι τέτοιο και θα έπρεπε να προχωρήσουμε και σε μια νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας. Υπήρξε συζήτηση με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, αλλά ενδιαμέσως υπήρξε και μία επιστολή που απεστάλλει από τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς που περιέχει και μία διευκρίνηση ότι εμείς ως Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων είμαστε η καθουσία αρμόδια επιτροπή, αλλά πρέπει η ΙΜΚΟ να εμπλακεί σε μια ενισχυμένη συνεργασία μαζί μας. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο τώρα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων στις βασικές υπηρεσίες με την κατάλληλη διαδικασία ρυθμιστικού χαρακτήρα στις τράπεζες, <clears throat> να υπάρχει υποχρέωση για όλες τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον γενικά για όλες τις τράπεζες, να μπορούν να παρέχουν βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι το χρήμα είναι ένα δημόσιο αγαθό όπως και να το αντιμετωπίσει κανείς και οι τράπεζες είναι ουσιαστικά διαχειριστές αυτού του δημοσίου αγαθού και ένας τραπεζικός λογαριασμός είναι απαραίτητο σε όλους για να μπορούν να λάβουν μέρος στην οικονομική ζωή. Επομένως θα πρέπει ο τραπεζικός λογαριασμός να είναι διαθέσιμος για όλους, είτε έχουν μια εργασία όπου έχει το μισθό τους, είτε είναι άνεργοι ή οτιδήποτε τέτοιο γιατί μπορούμε να πούμε ότι χωρίς ένα τραπεζικό λογαριασμό είναι κανείς χωρίς υπόσταση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον οικονομικό στίβο. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στο οικονομικό γίγνεσθε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υποχρεώσουμε τις τράπεζες να παρέχουν αυτές τις βασικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορούν να εξασφαλίσουν ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στο, σε ένα χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών. Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και σε μεταγενέστερα στάδια. Αλλά εγώ επιμένω ότι πρέπει να υπάρξει αυτό το καθήκον όλων των τραπεζών να θέτουν στη διάθεση όλων την ε, δυνατότητα αυτού του λογαριασμού και αυτό έχει και μια κοινωνική πολιτική, δηλαδή να μπορεί να βοηθήσει και ομάδες μειονεκτικές του πληθυσμού, όπως είναι μετανάστες, φοιτητές, άνεργοι κτλ. Ε, αυτό όπου πρέπει να υπάρχει, το σημείο αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει κάποια συμφωνία με την Κομισιόν για τα θέματα αυτά είναι το ποιε είναι οι ελάχιστε προποθέσει για να έχει κανεί τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα τραπεζικό λογαριασμό. Η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς κάτοικος που να είναι πολίτης της χώρας όπου ζητάει το τραπεζικό λογαριασμό, αλλά να είναι νόμιμα εγκατεστημένο στη χώρα αυτή. Αυτά λοιπόν για τις νομικές πτυχές. Προφανώς οικοθενοείται ότι πρέπει να υπάρξει και ισότητα ανταγωνισμού για όλες τις τράπεζες. Στην Ομοσπονδιακή Γερμανία υπάρχουν τράπεζες, κυρίως ταμιευτήρια που είναι υποχρεωμένες να δώσουν λογαριασμούς σε όλους και αυτό σημαίνει ότι υφίστανται πρόσθετο κόστος, ενώ άλλε τράπεζε μπορούν να μην το πράξουν αυτό. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλιστεί η ισότητα ανταγωνισμού μεταξύ όλων αυτών των τραπεζών. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν, όταν λέω γενικά πρέπει να ισχύει αυτό, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσει. Υπάρχουν σε ορισμένα κράτη οι λεγόμενες πιστοτικές ενώσεις που έχουν χαρακτήρα κλειστού, κλειστού τραπεζικού οργανισμού που δεν είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό και επομένως θα πρέπει να τύχουν κάποιες εξαίρεσεις από ένα τέτοιο κανονισμό. Πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν αυτό, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί ή όχι και μια άλλη μορφή εξαιρέσεως θα μπορούσε να αφορά για είδη τραπεζών τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν ιδιωτικούς λογαριασμούς και επομένως δεν πρέπει να τους επιβληθεί το άχθος να αποδέχονται λογαριασμούς για μεμονωμένα άτομα. Στο Βέλγιο υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει με αντισταθμιστικές πληρωμές όταν μια τράπεζα δεν συμμετέχει στην παροχή τραπεζικών λογαριασμών να μπορεί να αντισταθμίζει αυτό με κάποιες πληρωμές. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια ιδέα που θα μπορούσαμε να την λάβουμε υπόψη μας στη συζήτηση. Εγώ έχω συζητήσει με τραπεζικούς που μας είπαν ότι πάντα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αρνούνται την παροχή αυτών των ε, λογαριασμών. Στην Ομοσπονδιακή Γερμανία υπάρχει ένας κατάλογος που αναφέρει συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων έχει το δικαίωμα μια τράπεζα να αποκλείσει ένα πολίτη από την παροχή ενός τραπεζικού λογαριασμού. Θα μπορούσα να φανταστώ να μπορέσει να γίνει αυτό και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμως να προβάλλονται νομικά επιχειρήματα για να υπάρξει ένας τέτοιος κατάλογος, παραγωγός χάρη πολέμηση της ε, εγκληματικότητος, να αποφευθεί η έκπληση χρημάτων. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα σαφές νομικό εργαλείο. Ε, εάν δεν μπορεί λοιπόν μια τράπεζα ε, να δίνει σε όλους λογαριασμό χωρίς με τον τρόπο αυτό να ευνοεί ε, το πλήσιμο χρημάτων. Όταν λέμε βασικέ υπηρεσίε, μιλάμε για ένα βασικό λογαριασμό. Σε τι διαφέρει τώρα ένα βασικό λογαριασμό από άλλου λογαριασμού, Υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία μπορούμε να διατυπώσουμε και τα οποία παρουσιάζονται πολύ καλά στην πρόταση τη Κομισιόν, στη σύσταση τη ε, Κομισιόν. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένα λογαριασμό καταρχήν το γεγονό ότι μπορεί να πληρώσει χρήματα σε αυτόν τον λογαριασμό, να αποσύρει χρήματα από αυτόν τον λογαριασμό. Δεν είναι απαραίτητο να έχει τα στοιχεία του, να έχει τα λεγόμενα overdraft, δηλαδή να μπορεί κανείς να αποσύρει περισσότερα λεφτά από ό,τι περιέχει. Εγώ πιστεύω, και εδώ μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο για το θέμα αυτό, υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από την πλευρά των τραπεζών σε ό,τι αφορά την παροχή μιας ηλεκτρονικής κάρτας για να μπορεί ο κάθε πελάτης αυτόματα να αποσύρει χρήματα. Το πρόβλημα μιας τέτοιας κάρτας είναι πάντα ότι μερικές φορές υπάρχει καθυστέρηση στην ε, ε, στον καταλογισμό των αποσύρσεων που κάνει κάποιος με την κάρτα του από την τράπεζα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ελλείμματα στους λογαριασμούς το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε. Και ο βασικός αυτός λογαριασμός δεν θα πρέπει να συνδέεται με την υποχρέωση να αγοράσει ο πελάτης και άλλα προϊόντα σε μια τράπεζα. Γιατί πολλέ φορέ οι τράπεζε χρησιμοποιούν το βασικό λογαριασμό για να κάνουν προτάσει για περαιτέρω λογαριασμού, και αυτό πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι ο λαθασμένος δρόμος να ακολουθήσουμε. Ένα άλλο ερώτημα έχει να κάνει με μια προηγούμενη <clears throat> έκθεση για, τα, για τη δυνατότητα προσφυγής. Αυτό δεν συνδέεται απόλυτα με το θέμα της ε, χρηματοοικονομικής συμπερίληψης, το να μπορεί κανείς να προσφύγει σε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαμάχη. Το κόστος τώρα ενό τέτοιου, ενός τέτοιου βασικού λογαριασμού, και αυτό είναι σημαντικό, υπάρχει πάντα κάποιος κάποιο άχθος για ένα λογαριασμό. Οι τράπεζες είναι οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την κερδοφορία και αυτό το θέμα λοιπόν επομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. από μία πλευρά μπορεί κανείς να αιτιολογήσει ορισμένο, ορισμένες μορφές κόστους που επιβάλλονται στον πολίτη, στον καταναλωτή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς ένα βασικό λογαριασμό με έναν τρόπο ο οποίος ουσιαστικά δεν επιφέρει περαιτέρω κόστος στον χρήστη. Είτε λοιπόν είναι μηδενικό το κόστος ή αν θέσουμε ένα ανώτερο όριο στο κόστος ή αν προσανατολιστούμε προς το πραγματικό κόστος, όλα αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε κάποια ρύθμιση. Ένα τελευταίο στοιχείο είναι το, το θέμα της παροχής πληροφοριών και η ανάγκη εποπτείας αυτών των οργανισμών. Εδώ νομίζω μπορώ να παρακολουθήσω αυτά τα οποία λέει η σύσταση της Κομισιόν. Η Κομισιόν ζητάει από τα κράτη-μέλη να υπάρχει και μια ετήσια έκθεση για τα θέματα αυτά. Μια πληροφόρηση λοιπόν για τον αριθμό αυτών των βασικών λογαριασμών, πού βρίσκονται, σε ποιο πλαίσιο κτλ, πόσες αιτήσει έχουν γίνει για τέτοιους λογαριασμούς. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι έχει νόημα και για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας των Τραπεζών. Θα πρέπει και αυτή να πληροφορείται, αλλιώς δεν έχει πολυνόημα αυτή η ενέργεια και μπορούν πάντα να υπάρχουν, υπάρχουν και κάποιες περαιτέρω ενδείξεις και προτάσεις αυτά που λέει η Κομισιόν που εγώ δεν, τις, ε, δεν συμφωνώ απόλυτα όπως παραγωγός χάρη να λένε παραγωγός χάρη οι τράπεζες τους καταθέτες πόσο κοστίζει ο, ο κάθε λογαριασμός, η κάθε τραπεζική πράξη. Όλα αυτά είναι στοιχεία λοιπόν που εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το κ. Ζόνεφελ την Ορεστίνα έχουμε συζητήσει ήδη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν το ταχύτερο δυνατό μέσα στον επόμενο χρόνο να έχουμε ένα συγκεκριμένο έγγραφο εργασίας το ταχύτερο δυνατό γιατί στα μέσα του χρόνου η Κομισιόν θα ελέγξει και πάλι την σύστασή της και θα πρέπει μέχρι τότε η δική μας έκθεση να είναι έτοιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κλούτε και τότε δίνω το λόγο στους και εισηγητές. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Μίτσελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο επί του θέματος. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη λεπτομερέστατη έκθεση. Εδώ Στι λεπτομέρειες θα πρέπει να δώσουμε προσοχή, διότι λίγο πολύ εδώ θα επηρεαστούν οι επενδυτέ με χαμηλά εισοδήματα. Και εξαρτώνται πολλέ φορέ από την κοινωνική πρόνοια. Κατανοώ. Καταλαβαίνω των τραπεζών, αλλά οι τράπεζε περνάνε πολύ χρόνο έχοντα σαν στόχο του φοιτητέ, ξέροντα ότι κάποια στιγμή θα βγάλουν χρήματα οι φοιτητέ. Και πολλοί με χαμηλά εισοδήματα στο μέλλον θα βγάλουν και αυτοί λεφτά. Δεν θέλουν να έχουν για την υπόλοιπη ζωή τους χαμηλά εισοδήματα να είναι στην κοινωνική πρόνοια. Θα πρέπει να πιστούν ότι υπάρχουν καλές δυνατότητες και σε αυτό το τομέα οι τράπεζες. Και όσον αφορά το κόστος, το κόστος μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων ρευστών συνοδεία από αστυνομία και από στρατό και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεν είναι ίσονο σημασία θέματα είναι σχετικά θέματα και μπορούν να οικονομήσουν, ξεκονομήσουν χρήματα οι τράπεζε. Δεν ξέρω τι είναι σε άλλε χώρε, αλλά καλούνται να συμβάλλουν στη δική μου χώρα οι τράπεζε προ αυτό το κόστο. Κανεί δεν θα πρέπει να αποκλείεται από τραπεζικό λογαριασμό, εκτό ε, αν υπάρχουν κάποιοι πολύ σοβαροί λόγοι για τέτοιο, για αποκλεισμό. Κανεί δεν θα πρέπει όμω να υποχρεούται να έχει τραπεζικό λογαριασμό. Το Ιρλανδικό Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε μια έκθεση για μια στρατηγική για την οικονομική ένταξη το 2011 και κατέληξε σε διάφορα συμπεράσματα. Ένα από αυτά ήταν ότι ε, μέσω τραπεζικού λογαριασμού καταβάλλονται οι διάφορες κοινωνικές εισφορές είναι ο καλύτερο τρόπος για την, α, ε, ε, το να, να όχι να εκμεταλλεύονται, να, να, να, καλύπτονται από αυτή την κοινωνική ασφάλιση αυτοί που έχουν χαμηλό εισόδημα. Χρειάζονται σωστέ διευθετήσει για να λειτουργήσει το σύστημα. Προσβλέπω ε, το ταχύτερο δυνατό να παραλάβω την έκθεση αρχές του νέου έτους αλλά θα έλεγα στον εισηγητή ότι η γενική εικόνα, το πλαίσιο ε, είναι αποδεκτό. Πρέπει να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες, διότι εκεί κρύβεται και ο διάβολος, τις λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να ανησυχούμε υπερβολικά για το κόστος που πρέπει να υπομειστεί η τράπεζα έχει και πολλά φέλη τράπεζα όταν έχει λογαριασμό και παίρνουν χρήματα από το λογαριασμό. Και όλοι οι αποδέκτες διαφόρων τη ε, της κοινωνικής πρόνοιας επειδή ζουν συνήθως ε, με χαμηλό κόστο ε, κόστος μένουν κάποια χρήματα στο λογαριασμό τους ε, υπάρχουν και συν και πλήν, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ένας τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να διαθέσει μόνος για οποιονδήποτε το επιθυμεί, σχεδόν κανείς να μην αποκλείεται, αλλά να μην υποχρεούται κάποιο να έχει λογαριασμό. Έκανε καλή προετοιμασία ο εισηγητή και εν αυτό το χρόνο θα υποβάλω και εγώ τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ. Ο κύριο Λούτφιξον είναι εδώ. Α, ναι, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Εδώ θέλουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή με θετικό πνεύμα και για αυτό το ζήτημα. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλά εργαλεία για να επιφέρουμε μεγάλες βελτιώσεις για ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών. Από τη δική μου τη σκοπιά και μακροπρόθεσμα είναι απολύτως εφικτό να έχουμε και περιορισμένη και ισόρροπη νομοθεσία που ταυτόχρονα θα ενοποιεί την εσωτερική αγορά για τη διασυνοριακή κινητικότητα, την ψηφιακή ανάπτυξη, την, ε, τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα πρέπει να καλυφθεί η ιδέα ότι θα έχουμε εδώ νομοθεσία και σχετικούς κανονισμούς που να προκύπτει από το έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο θα πρέπει να εκλειφθεί ως σημείο αφετηρίας. Δύο ζητήματα πρέπει να έχουμε κατά νου συνεχώς. Πρώτα απ' όλα ότι ωφέλη θα προκύψουν εάν το σύστημα είναι γενικευμένο και όσο το δυνατόν καθολικότερο, ώστε όλες οι τράπεζες να έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν ένα οπλοστάσιο, μια ολόκληρη πανοπλία παρέτρα μάλλον, συγγνώμη, από βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε και τον κοινωνικό στιγματισμό που μπορεί να προκύψει εάν ε, μόνο κάποιες τράπεζες ε, παρέχουν τη δυνατότητα τέτοιου είδους ε, τραπεζικών λογαριασμών. Πρέπει όλοι οι πολίτες, σε όλους τους, τρο... τους τραπεζικούς, να καλύπτονται, διότι δεν θα πρέπει μόνο ορισμένοι να έχουν πρόσβαση σε ειδική κατηγορία λογαριασμών. Δεν θέλουμε λοιπόν μόνο για μια μικρή ομάδα πολιτών κοινωνικά ωφέλη. Επίσης, υπάρχουν βασικές αρχές ό,τι αφορά τον καθορισμό των τιμών και του κόστους. Οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες σίγουρα θα εξαρτηθούν πολύ και από τη σχέση τιμής και κόστους. Για αυτούς που συχνά αποφεύγουν τις τράπεζες, πολλές φορές το κάνουν αυτό και λόγω του κόστους. κάποιοι περιμένουν αρκετά μέχρι να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, διότι δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος. Πολλές φορές φτάνει και τα 10 ευρώ για να κλέωσαν το λογαριασμό από συγκεκριμένη πηγή. Πρέπει λοιπόν να δούμε εδώ ποιο σύστημα θα λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει διάφορα κριτήρια. Εδώ τα κράτη-μέλη αναφέρουν ε, διάφορα εδώ μάλλον αναφέρονται διάφορα στοιχεία για τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Η νομοθεσία στον τομέα αυτό θα πρέπει να συμβάλλει ώστε να αναπτυχθεί η ψηφιακή ατζέντα όλοι οι πολίτες, ακόμη και εκείνοι που θεωρούνται λιγότερο ελκυστικοί για τις τράπεζες, θα πρέπει να αξιοποιούν τις δυνατότητες από τις νέες εξελίξεις. Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου θα πρέπει να γίνουν ε, μια συνήθεια για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε εδώ ε, σημάδια ότι θα υπάρξει μια πορεία αρκετά μακρά μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Οι τραπεζικέ υπηρεσίε στο διαδίκτυο συχνά είναι φτηνότερε. Όμω είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση για ορισμένε ομάδε των πολιτών. Και μάλιστα οι τράπεζε του θεωρούν και προβληματικέ ομάδε. Εδώ οι τράπεζε τείνουν να είναι κάπω ε, αυστηρέ. Οι τραπέζι συναλλαγέ στο διαδίκτυο είναι απλέ, όμω Θα πρέπει να έχουμε υπόψη κάποιες ομάδες του πληθυσμού ως στόχους. Τα πράγματα πρέπει να απλοποιηθούν και για τους πελάτες και για τις τράπεζε. Θα πρέπει λοιπόν, ελπίζω, μάλλον η συνεργασία μας τις επόμενες ε, εβδομάδες και μήνες να είναι επικοδομητική και να καταλήξουμε σε μια καλή λύση, ώστε να συμφωνήσουμε σε λογικέ βάσει. Ευχαριστούμε κυρία Γκουλάρ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ εξ ονόματος του Φιλίπ Τεμπακέρ που είναι ο σκιώδης μας συγητής, εκφράσω την άποψη των φιλελευθέρων και με την ευκαιρία αυτή δίνω και τη δική μου γνώμη γιατί είμαι αντιπρόεδρος της ε, διαπρακταξιακής ομάδος που προεδρεύεται από τον Νίκο Μεντεστεβίγκο κατά της ένδυας. Είναι μια δράση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ένδυας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κινητοποιημένοι για τα θέματα αυτά. Και μίλησα ήδη με τον ε, Γιούργεν Κλούτε Θέλουμε όλοι να προχωρήσουν τα πράγματα αυτά. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν γερθεί. Το θέμα του κατά πόσον συγκεκριμένα μπορούμε να περιοριστούμε, να έχουμε μια σύσταση η οποία δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να προχωρήσουμε να περάσουμε και επέκεινα αυτού του πλαισίου. Είναι καλύτερα να έχουμε ένα στενό αλλά δεσμευτικό πλαίσιο παρά να αφήσουμε τις χώρες μέλη να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό. Επίσης πρέπει να είναι σαφές να αποφασίσουμε αν πρέπει να είναι εγκάρσια αυτή η υποχρέωση να υπάρχει μονάχα ένας πάροχος τέτοιων λογαριασμών. Εγώ νομίζω ότι αυτή η υποχρέωση μπορεί να αφορά πάρα πολλά άτομα. Γιατί λοιπόν μόνο μία τράπεζα και όχι πολλές. Πώς θα εξασφαλίσουμε τις, ναι, τις σωστές ανταγωνισμού και πώς θα εξασφαλίσουμε και την ισορροπία σε γεωγραφικό επίπεδο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πραγματικά με μεγάλες συγκεντρώσει πληθυσμού που ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο θα πρέπει να εστιάσουμε στα πραγματιστικά και όχι στα αφηρημένα θέματα. Γι' αυτό η διαπαραταξιακή ομάδα κατά της ένδυας θα συναντηθεί του χρόνου με εκπροσώπους αυτών που έχουν δυσκολία για να έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς για να ακούσουμε και τις δικές τους απόψεις, ποιες είναι οι πραγματιστικές λύσεις που προτιμούν αυτοί οι ίδιοι. Και επίσης πρέπει να ξέρουμε σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα γίνουν όλα αυτά Κατά την άποψή μου είναι εκατομμύρια ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και επειδή κάθε μέρα ακούνε όλοι αυτοί να μιλάνε για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το χρηματοπιστωτικό τομέα, ίσως το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ασκήσει κάποια πίεση προς τις τράπεζες, χωρίς υπερβολή, για να μπορέσουν και αυτοί να συμβάλλουν ως τραπεζικός τομέας στο να υπάρξει η κοινωνική δικαιοσύνη στις χώρες μας. Θέλω να κλείσω με μια μικρή σημείωση γιατί πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Εφέτος, και δεν είναι τυχαίο, το business book του χρόνου των Financial Times και της Goldman Sachs δόθηκε σε δύο οικονομολόγους της Ηνωμένες Πολιτείες στο MIT, η Εστέντη Φλός, μια Γαλλίδα και ένας κύριος από την Ινδία και δεν θέλω να δολοφονήσω το όνομά του, αλλά η ιδέα ήταν ότι εξέδωσαν ένα βιβλίο που λέγεται Poor Economics και που τονίζει πως θα πρέπει η βοήθεια προς φτωχότερους να σχεδιαστεί με τη δική του συμμετοχή και ότι αυτοί πράγματι συμβάλλουν στην κοινωνία. Αν τους αφήσουμε στην άκρη του δρόμου, χάνει όλη η κοινωνία και όχι μόνο αυτήν. Εάν ακόμα και η Goldman Sachs και οι Financial Times θέλουν να υποστηρίξουν αυτό το βιβλίο, ίσως και το δικό μας κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ένα πιο κομβικό ρόλο για να υποστηρίξει τα άτομα τα οποία πλήττονται από την ένδια. Νομίζω λοιπόν ότι είμαι απόλυτα για τα, ανοιχτή για τα θέματα αυτά, το ίδιο και ο Φιλίπ Τεμπάκερ και σας τονίζω και πάλι ότι έχουμε μια ευκαιρία να δώσουμε το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν είναι μονάχα για τους λεφτάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι σκιώδη συζητητή για την ομάδα μου, αλλά έρχομαι σε επαφή διάφορε οργανώσει. Εργάζομαι με διάφορου οργανισμού, διάφορου φορεί στην εκλογική μου περιφέρεια για να δούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση των φτωχών στι χρηματοστατικέ υπηρεσίε και συζήτησα πολύ με διάφορου φορεί ε, πιστοτικούς και προσπαθούμε να βρούμε προγράμματα για να βοηθήσουμε του ανέργου να έχουν πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση και να ξεκινήσουν δικέ του επιχειρήσεις. Όταν είδα ότι αυτό το θέμα ήταν στην ημερήσια διάταξη θεώρησα ότι θα ήταν σημαντικό να ακούσω τι απόψει που θα εκφραζόταν. Δύο βασικά σημεία έχω να τονίσω. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικότατοι όπως είπε και η κυρία Γκουλάρ να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να είμαστε σίγουροι ότι όταν θα έχουμε πολιτικέ που έχουν στόχο του λιγότερο τυχερού από εμά ή του φτωχότερου από εμά, να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε να δούμε και ποιε θα πετυχαίνουμε αυτά που θέλουμε. Να μην έχουμε ε, κάποιε συνέπειε που δεν θέλουμε. Ε, Όμω στο subprime, στην κρίση του subprime τελικά ήταν επειδή δόθηκαν δάνεια σε ανθρώπου που δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν. Και είχε ε, οδήγησε στην κρίση τη γνωστή των subprimes δεν μιλάμε για δάνεια όμως εδώ, μιλάμε για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Και κάτι άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός στις τράπεζες, έναντι τραπεζών. Γιατί το λέω αυτό. Ίσως λησμονούμε τον ζωτικό ρόλο που οι διάφορες ασφαλιστικές παίζουν ρόλο. Διάφοροι φορείς ασφάλισης και διάφοροι άλλοι φορείς συνεταιριστικοί που δανείζουν χρήματα και έχουν μέλη θα πρέπει να γνωρίσουμε το ρόλο που παίζουν και αυτοί. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις συνέπειες και να δούμε εάν πούμε στις τράπεζες ότι θα πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες που είναι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες μήπως με τη μία ε, δημιουργούμε πρώτα απ' όλα θέλω να το κάνουν αυτό οι τράπεζες αυτό είναι άσχετο ίσως δεύτερον μήπως ασκούμε πιέσεις σε εκείνους που παρέχουν τις υπηρεσίες που δεν είναι τράπεζες και παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες οικονομικές στους στοχούς. Εάν η συνέπεια αυτού που κάνουμε είναι να βγάλουμε εκτός τους άλλους φορείς, συνεταιριστικούς και ασφαλιστικούς φορείς, διότι χάνουν χάνουν των τραπεζών, δεν το θέλουμε αυτό. Μάλλον δεν κινούμαστε προς τα εκεί, αλλά το λέω για να προσέξουμε πάρα πολύ τι κάνουμε. Και δεν θα πρέπει να ξεγελιόμαστε. Ε, θεωρούν ότι ε, βάζουν στις, σε, από ταμευτικό λογαριασμό ε, και κρατάνε σαν απόθεμα τα χρήματα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε ε, τους στοχούς. Ε, δεν τα αφήσουν σε κατάθεση ε, απλή, τα, βάζουν σε, τα κλείνουν σε λογαριασμούς. Δανείζεις χρήματα σε τράπεζες. Δεν τα βάζεις σε ταμιευτήριο. Και αυτό είναι το πρόβλημα του τραπεζικού τομέα εν γέννη. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ειλικρίνεια όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση των φτωχών στι τραπεζικέ υπηρεσίε, αλλά δεν απαραίτητο αυτέ οι υπηρεσίε οι οικονομικέ και χρηματοπιστωτικέ να προέρχονται απαραίτητα από τι τράπεζε. Ευχαριστώ κύριε Καμάλο. Ο κύριο Γιγκό. έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα εγώ χαίρομαι και το γεγονός ότι συζητούμε τα θέματα αυτής της έκθεσης τώρα είναι σημαντικό να θυμηθούμε όλοι πώς φτάσαμε εδώ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Εγώ θυμάμαι τη συζήτηση που κάναμε ως συντονιστές για το θέμα αυτό. Και ήταν πριν από πολύ καιρό που ο Γιούργεν πήρε την εντολή να αναλάβει την εισηγεσία αυτής της έκθεσης. Ότι τώρα έχουμε φτάσει στο επίπεδο μιας έκθεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας εφόσον παίρνουμε πολλές ε, πρωτοβουλίες από την Κομισιόν, δεν χρειάζεται να κάνουμε πρόσθετες εκθέσεις πρωτοβουλίας. Αλλά το γεγονός ότι κάνουμε κάτι τέτοιο εδώ δεν γίνεται τυχαία. Γίνεται γιατί αυτό ήταν ένα κομμάτι του σχεδίου εργασίας της Κομισιόν και η Κομισιόν δεν μας έχει δώσει μια νομοθετική πρόταση στα θέματα αυτά. Προχώρησε μονάχα προς μια σύσταση προς τα κράτη-μέλη. Βλέπω τους εκπροσώπους κομισιών, οι οποίοι βέβαια δεν είναι οι υπέτειοι για κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να ξέρουν όμως το εξής, επειδή εγώ έκανα κάποια έρευνα στα θέματα αυτά, να θυμούνται πώς φτάσαμε εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πω αυτό δημόσια. Η ιστορία είναι, και εδώ υπάρχει και μια φήμη που θα ήθελα να την αρνηθείτε ή να την επικυρώσετε, πήρα άκουσα από έγκυρες πηγές την εξής εξήγηση. Έλαβε χώρα μια συνάντηση υψηλού επίπεδου μεταξύ των ε, ηγετών <clears throat> της ε, Κομισιόν και των εκπροσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου και υπήρξε μια αίτηση να μειωθεί η επίπτωση της, ε, των νέων ρυθμίσεων και ακριβώς το θύμα αυτής της νέας πορείας ήταν η οδηγία αυτή για τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτό είναι μια ηρωνία. Γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και αυτό ήταν, όπως είπατε, το τμήμα του πακέτου που αφορούσε τους ασθενέστερους και τους ενδέστερους ώστε θα είχαν έτσι κάποιο πλεονέκτημα μετά από όλα τα μειονεκτήματα που δημιούργησε για όλους μας η χρηματοπιστωτική κρίση. Είναι κρίμα λοιπόν το γεγονός ότι δεν μπορούμε πια να διαπραγματευτούμε για την διατύπωση μια οδηγία και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτό το εργαλείο. Αυτό δείχνει όμω και την ισχύ του Κοινοβουλίου. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι εξουσίε που έχουμε βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. σω πρέπει να το πράττουμε πιο συχνά. Είναι πολύ θετικό ότι προχωρούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε προσεκτικοί. Και τώρα μιλάω για την ουσία. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία και συνένεση, αλλά υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να μην δημιουργήσουμε λοιπόν <clears throat> ένα ειδικό χρηματοπιστωτικό τομέα ο οποίος συνδέεται μόνο με το να είναι υπηρεσίες χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα για τους φτωχούς. Γιατί με τον τρόπο αυτό απλώς αναπαράγουμε μια νέα μορφή διακρίσεων η οποία <clears throat> θα μπορεί να φέρεται από το χαρακτηριστικό κώδικα της κάθε τράπεζας. Αυτό θα ήταν αρνητικό. Δημιουργήθηκαν φορείς για να καλυφθεί αυτό το κενό το οποίο έχει αφαιθεί από τις λεγόμενες κύριες τράπεζες και τα ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αλλά μίλησα και με τους εκπροσώπους των πιστοτικών ενώσεων. Είπαν όχι, δεν θέλουμε οι άλλες τράπεζες να αποκλείσουν τους καταναλωτές μας και τους καταθέτες μας. Δεν θέλουμε να σταματήσει αυτή η νομοθεσία γιατί ξέρουν ότι αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν καλύτερα είναι η δανειοδότηση των φτωχότερων στην κοινωνία μας. Δεν μπορείτε να υποχρεώσετε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία να είναι καλή ως δανειστής των πιο φτωχών. Δεν είναι η δουλειά τους, δεν τους ενδιαφέρει, δεν θα το κάνουν. Μπορούμε όμως να τους υποχρεώσουμε να προσθέσουν σε όλους ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό, γιατί δεν θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι ο τομέας αυτός των πιστοτικών ενώσεων δεν θεωρεί δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι θα πρέπει να ξεκολουθήσουν να δρουν διακριτικά κατά των φτωχών. Δεν λοιπόν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να θυμόσαστε ότι οι πιστοτικέ ενώσει έχουν σαν κύριο στόχο να βοηθήσουν του ανθρώπου και όχι να έχουν κερδοφορία. Τι θα έφερε τώρα μια οδηγία στα θέματα αυτά, θα βοηθούσε να σταματήσει αυτή η συνεχής σπήλωση και διάκριση που υπάρχει σε πολλά κράτη-μέλη. Όταν σπούδαζα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θυμάμαι κάποιες επιστημονικές μελέτες που έδειχναν ότι υπάρχουν περιοχές όπου ζουν περισσότεροι φτωχοί <clears throat> και όπου ορισμένες ε, τράπεζες δεν ανοίγουν υποκαταστήματα σε αυτές τις περιοχές για λόγους αρχή. Αυτό είναι λοιπόν μια κατάσταση που παρατηρείται και στη Γερμανία. Δεν θέλω λοιπόν να ισχύσει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό υποστηρίζω τη γενική κατεύθυνση αυτής τη έκθεσης και χαίρομαι και για την ιδέα να έχουμε περιορισμένα αλλά δεσμευτικά κριτήρια. Αυτό είναι πάρα πολύ θετική ιδέα για μένα και ελπίζω ότι αυτή η, νομοθετική, η έκθεση νομοθετική πρωτοβουλίας μπορεί να μας βοηθήσει και την Κομισιόν και το Συμβουλίο ακόμα να έχουν μια πιο επικοδομητική προσέγγιση Ξέρω ότι υπήρχαν νομικά επιχειρήματα που βασίζονται στην επικουρικότητα εναντίον μιας τέτοιας ε, ρύθμισης, αλλά αυτό δεν είναι <clears throat> ιδιαίτερα πιστικό γιατί και σε άλλους τομείς προχωρούμε σε κοινά πρότυπα για τις υπηρεσίες, όπως παραδείγματος το δικαίωμα για ευρυζωνική υψηλή ταχύτητα πρόσβαση στο ίντερνετ, όπου θέλουμε να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Λοιπόν, γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για τους τραπεζικούς λογαριασμούς συμφωνώ ότι αυτό τελικά θα είναι και προς το συμφέρον του χρηματοπιστωτικού τομέα και γι' αυτό προσβλέπω <clears throat> στη συνεργασία με τους άλλους συζητητές για το θέμα αυτό και ελπίζω ότι σύντομα θα μπορούμε να έχουμε μια πραγματική νομοθετική έκθεση και θα ξεπεράσουμε απλώ το επίπεδο μιας έκθεσης πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου. Και αυτό θα είναι ένα καλό χριστιογεννιάτικο δώρο και αναρωτιέμαι αν θα μπορούσατε να δώσετε το λόγο και στην Κομισιόν για να ακούσουμε ποια είναι η δική τους θέση, τι προβλέπουν να κάνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σύστασης τους προς τα κράτη-μέλη, αν θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στεναρή δράση από την πλευρά των κρατών μελών και δεν χρειάζεται να υπάρξει περαιτέρω δράση από αυτούς. Εγώ μέχρι τώρα πάντως δεν έχω δει καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε κάποιες θετικές ιστορίες επιτυχίας από την Κομισιόν πριν από τα Χριστούγεννα. Ενδιαφέρομαι λοιπόν να ξέρω αν είσαστε ήδη προετοιμασμένοι να προχωρήσετε προς μια νομοθετική δράση εάν τα κράτη-μέλη δεν ανταποκριθούν στη σύστασή σας. Ευχαριστούμε κύριε Γκόλντ. Θα ζητήσω και από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο, όμως και εγώ θέλω κάτι να τονίσω. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των προτύπων της ίδιας διακρατικής τράπεζας που λειτουργεί εντός μιας χώρας ή και σε μια άλλη. Να σας πω τι συμβαίνει σε μένα, στη δική μου χώρα. δεν υπήρχαν τραπεζικές υπηρεσίες για τους πολίτες, τραπεζικοί λογαριασμοί. Η πρώτη τραπεζική δραστηριότητα που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια ήταν να ξεκινήσουν να ανοίγονται τραπεζικοί λογαριασμοί για να λαμβάνουν οι πολίτες τους μισθούς τους. Έτσι ανακαλύψαμε, βάζοντας λεφτά στους λογαριασμούς, ότι μπορούμε να λάβουμε εκεί την αμοιβή, το μισθό μας, και ότι έπρεπε παρόλα αυτά να καταβάλουμε κάποιο τέλο για, για κάθε συναλλαγή που γινόταν στον τρέχοντα λογαριασμό. Νομίζω και ξέρω ότι σε άλλε χώρε τέτοια τέλη δεν υπάρχουν. για την κίνηση των χρημάτων από τον τρέχοντα λογαριασμό, αλλά αυτό είναι κατάχρηση των δυνατοτήτων που έχουν οι τράπεζες για να αντλούν χρήματα από τι συναλλαγέ των πολιτών. Τώρα, αν δεν, δεν σα πειράζει, κύριε Κλούτε, αυτό να το έχετε κατά νου, συντάσσοντα την έκθεσή σα. Να υπάρχει και δικαιοσύνη στον τραπεζικό τομέα, στι τραπεζικέ υπηρεσίε για, όλους, για όλε τι χώρε. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει από του βουλευτέ, να ζητήσω από τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το όλο θέμα που βρίσκεται και στο κέντρο των προβληματισμών του Επιτρόπου, του κ. Μπαρνιέ. Ελπίζουμε η έκθεση αυτή πρωτοβουλία να είναι έτοιμη σύντομα. Και μάλιστα ταυτόχρονα με την έκθεση που πρέπει να ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ερχόμενο καλοκαίρι. Δυστυχώ, κύριε Γκίγκολ, δεν έχω καλά νέα για τα Χριστούγεννα για εσά. Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από τα κράτη-μέλη που υποτίθεται ότι πρέπει να μα ενημερώσουν ω το τέλο του Ιανουαρίου. <coughs> Έξι μήνε μετά τη δημοσίευση τη ε, σύσταση. Εδώ δεν έχουμε λάβει ακόμη τίποτα. Βεβαίω, ε, ξέρουμε ότι συστήματα ανάλογα υπήρχαν ήδη σε κάποια κράτη-μέλη, είτε από πρόνοια των ρυθμιστικών αρχών, είτε με την αυτορύθμιση. Αλλά άλλε πληροφορίε από τα κράτη-μέλη δεν έχουμε ως προς την συνέχεια που είχαν σκοπό να δώσουν στη σύσταση αυτή. Να σας καθησυχάσω πάντως, εάν φανεί ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο αυτής της σύστασης είναι ανεπαρκή, τότε θα αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μπανιά νομίζω υπήρξε πολύ κατηγορηματικό όπω το θέμα αυτό, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι ο κάθε Ευρωπαίο πολίτη που κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πρόσβαση σε έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Και το θέμα λοιπόν τη οικονομική συμμετοχή, τη χρηματοπιστωτική αυτή συμμετοχή. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε και από ένα μέλο τη Επιτροπή σα, εδώ προστίθεται η πρόσβαση των ε, μη κατοίκων στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό παραπώνων από τους Ευρωπαίους πολίτες που δεν είναι κάτοικοι συγκεκριμένου κράτους μέλους και τους αρνούνται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο κράτος μέλους. Αυτό είναι κάτι που καλύπτεται από τη σύσταση, αλλά επιπλέον θα πρέπει να καλύπτεται και από κάθε μελλοντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμμεριζόμαστε ένα μεγάλο αριθμό της παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον εισηγητή Κλούτε, η ροή του ρευστού, τα τέλη των, για τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς θα πρέπει να είναι λογικά, ανάγκη να προβλεφθούν και ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, καινοτόμα, σύγχρονα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σύστασή ήθελε να αφήσει και ένα περιθώριο ευελιξία στα κατημέλια προ του στόχου του. Να μην υποχρεώνει το σύνολο των τραπεζών να παρέχουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό, απλώ να είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε θα ισχύει. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε να έχουν πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Λόγω χάρη στη Γαλλία, εφόσον είναι αναγκαίο, με τον διορισμό κάποια κεντρική αρχή, όπω στη Γαλλία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ας... Αυτή, είναι αυτή η τράπεζα που παρέχει το βασικό τραπεζικό λογαριασμό σε κάποιον Γάλλο πολίτη πω, εφόσον άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του αρνήθηκε την πρόσβαση. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε κάποιο περιθώριο ευελιξίας και στα κάτι μέλη, γιατί υπάρχουν διαφορετικά συστήματα και αυτό που για μας είναι σημαντικό ήταν ο τελικός στόχος να διαθέτουν όλοι οι πολίτες που το επιθυμούν έναν τραπεζικό λογαριασμό, έστω βασικό. Αυτό αφήνει κάποια ευελιξία και στα χρηματοπιστωτικούς στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στα trading unions και νομίζω ότι τον τελικό λόγο θα πρέπει να τον έχουν σε κάθε περίπτωση εδώ τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ λοιπόν, θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή και με το Ευρωκοινοβούλιο για την προετοιμασία αυτής της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας η οποία οπωσδήποτε θα συμβάλλει στην προετοιμασία πρόσθετων πρωτοβουλίων, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ερχόμενο Ιούλιο πρέπει να δημοσιεύσει ε, σχετικά αποτελέσματα και δούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν τα όσα πρέπει η σύσταση του περασμένου Ιουλίου. Ευχαριστούμε. Κύριε Κλούτε, θέλετε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις που διατυπώθηκαν. Υπάρχει περισσότερη συνένεση από ό,τι προσδοκούσα και αυτό θα διευκολύνει το έργο μου. Στον κύριο Καμάλ ήθελα να πω ότι ότι οι πιστοτικές ενώσεις, credit unions, είναι διαφορετικές καταστάσεις από τις γενικές τράπεζες και υπάρχουν και άλλες μορφές όπως οι συνεταιριστικές τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε στην ε, Γερμανία συνεταιριστικές τράπεζες που δίνουν λογαριασμούς για όλους αυτούς οι οποίοι το επιθυμούν και είναι μέλη της Ένωσης. Επίσης υπάρχει το θέμα των μικροπιστώσεων που αντιμετωπίσαμε και στην ακρόαση που κάναμε νωρίτερα μέσα στον ε, χρόνο αυτό το 2011. Ακούσαμε πολλές φορές από αυτούς οι οποίοι έλαβαν ε, μέρος σε αυτές τις ακροάσεις για τις μικροπιστώσεις και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και δεν θα είχε νόημα να συνδέσουμε τις μικροπιστώσεις που αφορούν άτομα σε μεγάλη δυσκολία με λογαριασμούς οι οποίοι αφορούν πάλι όλους τους πολίτες. Θα πρέπει να κρατήσουμε χωριστά αυτά τα θέματα και μου φαίνεται λογικό να παραμείνουμε μόνο στα πλαίσια της συγκεκριμένη εντολής που έχουμε. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω αν υπάρχουν συγκεκριμένες αιτήσει για τα θέματα αυτά. Και κατά τα άλλα, καλό βράδυ σε όλους, θα συνεχίσει η εργασία μας και έχουμε ακόμα δρόμο να διατρέξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Τελειώνει λοιπόν η συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας είναι στις 9 Ιανουαρίου και σας εύχομαι σε όλους καλές γιορτές. you